We would like to, to start the meeting. Good afternoon, everybody. We have a very heavy agenda for this Γεια σας, έχουμε μια πολύ βαριά ημέρα διάταξη σήμερα το απόγευμα. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε για να μπορούμε να είμαστε σε θέση να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις που έχουμε σήμερα το απόγευμα σε σχέση με τους ομιλητές, σε σχέση με τα ερωτήματα, αλλά και τις απαντήσεις. Αγαπητά μέλη, ομιλητές, συμμετέχοντες, σας καλωσορίζω στη δημόσια ακρόαση για την Στατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συμπερίληψη στο Ρωμά. Οργανώνεται από την Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πλαίσια μιας έκθεσης. Η κυρία Λίδια Γιαρόκα είναι η συγγετρία για αυτή την έκθεση. Και έχουμε την ε, Επιτροπή μας, η οποία έχει Συγχρόνω και τη συμμετοχή της Επιτροπής Απασχόλησης μέσα στα πλαίσια του άρθρου 50 του κανονισμού μας. Θέλω επίσης να χαιρετήσω και την κυρία Κίνγκα Γκόλ, η οποία είναι συντάκτρια γνωμοδότης Επιτροπής Απασχόλησης, ο κύριος Στάκουλα από την Επιτροπή ε, Πολιτισμού και επίσης και ο κύριος Κόβατσεφ από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ως συζητητή γνωμοδότηση. Έχουμε πολλούς ε, ομιλητές οι οποίοι είναι καλεσμένοι μας, την κυρία Ρέντινγκ, η οποία είναι η επίτροπος αρμόδια για τα θέματα αυτά. Έχουμε εκπροσώπους της Ουγγρικής και της Βελγικής Προεδρίας και διακεκριμένους καλεσμένους από την κοινωνία των πολιτών. Έχουμε επίσης καλεσμένους από το Συμβούλιο της Ευρώπης μία πλειάδα αποκαλεσμένους που καλύπτουν το φάσμα ενδιαφέροντος. Το πρόσφατο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενεκρίθη στις 9 Σεπτεμβρίου 2010 σε σχέση με την κατάσταση των Ρώμα και την ελευθερία διακίνησή τους και αντιμετωπίστηκε με μεγάλη ε, κοινή ευθύνη, κοινό αίσθημα ευθύνης από τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ομοφωνία. Είναι μια ευκαιρία επίση να δώσουμε κάποια ανάδραση για τα συμπεράσματα τη δεύτερη Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Κορυφή για την συμπερίληψη στο Ρωμά, που είναι στην ε, Κόρντοα 8 και 9 Απριλίου 2010 και έχει σαν στόχο να ενισχύσει τη διαθεσμική συνεργασία και να ξεκινήσει ένα επικοδομητικό διάλογο με την κοινωνία των πολιτών. Η ακρόαση μα θα δώσει στην Κομισιόν την ευκαιρία να παρουσιάσει στο Κοινοβούλιο και στο Γενικό Κοινό τη σκέψη τη για τα θέματα αυτά που θα αποτελέσουν και τη βάση για την έκθεση της ε, ειδική μονάδας για τους Ρωμά που προβλέπεται να δημοσιευθεί με στους επόμενους δύο μήνες. Η δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαιώνεται και από το μεγάλο ενδιαφέρον της τωρινής Βελικής Προεδρίας και θα είναι φυσικά και μία από τις προτεραιότητες της επικείμενης Ουγγρικής Προεδρίας η οποία προβλέπει να θέσει το θέμα της συμπερίληψης των Ρωμά ως ένα από τα ζητήματα προτεραιότητα τη προεδρία τη. Η επιτυχία μια τέτοια στρατηγική εξαρτάται από τη συμμετοχή τη κοινωνία των πολιτών και από τη συμμετοχή όλων των φορέων που είναι ενεργοί στον τομέα αυτό και έχουν ιδιαίτερη εμπειρία για τα θέματα αυτά και επομένω μπορούν να μα δώσουν την εμπειρογνωμοσύνη του. Αυτό είναι και το πλαίσιο μέσα στο οποίο συνεχίζουμε την εργασία μα για την έκθεση πρωτοβουλία αυτή. Νομίζω ποτέ στο παρελθόν μια έκθεση πρωτοβουλία δεν θα μπορούσε να έχει τόσο μεγάλη επιρροή στις κεντρικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η έκθεση και το περιεχόμενό της, που ελπίζουμε ότι θα εγκριθεί σύντομα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε τρία τμήματα της ακρόασης. Το πρώτο αφορά τις απόψεις των ευρωπαϊκών θεσμών και θα έχουμε φυσικά την κυρία Ρέντινγκ, η οποία θα λάβει τον λόγο εξώματος της Επιτροπής η δεύτερη, το δεύτερο τμήμα θα αφορά τον ε, φορέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, το Συμβούλιο της Ευρώπης και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Και αύριο έχουμε την τρίτη, το τρίτο τμήμα με τον κύριο Λάσο Άντορ, ο οποίος είναι ο Επίτροπος Απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέσεων και Συμπερίληψης και θα ακούσουμε τις απόψεις πολλών φορέων που αντιμετωπίζουν τα θέματα αυτά το πρόγραμμα ανάπτυξη των ΗΠΑ, Εθνών και φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όποιος θέλει να λάβει το λόγο θα πρέπει να το αναφέρει στο Προεδρείο λέγοντας ποιο είναι το όνομά τους και ο φορέας τους και αυτό με ένα ειδικό έντυπο το οποίο θα κυκλοφορήσει σε όλους. Θα δώσω καταρχήν το λόγο στην κυρία Μπέρες, εξ ονόματος Επιτροπής ε, Απασχόλησης και Κοινωνικών Θεμάτων και μετά θα ζητήσω από την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, την κυρία Ρέντινγκ, να λάβει το λόγο αμέσως μετά, γιατί μετά γιατί έχει και άλλε υποχρεώσει σήμερα και δεν θα μπορέσει να μείνει όλο το διάστημα αυτό. Κυρία Μπέρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, δεύτερη φορά στο, στην περίοδο αυτή του Κοινοβουλίου ασχολούμαστε με του ΡΟΜ. Ε, οι δύο επίτροπέ ε, βρίσκονται εκ των πραγμάτων σε μια ακρόαση Τη μια φορά ήταν μετά από τις δηλώσεις με πολύ κουράγιο της Επιτρόπου κύρια Ρέντινγκ που επιτρέψα να περάσουμε σε ένα καινούριο στάδιο για να αναλάβει αυτό το θέμα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαίρομαι λοιπόν μετά από όλη αυτή την κατάσταση που βλέπω την αποφασιστικότητα του Προέδρου του Κοινοβουλίου, του κ. Μπούζεκ, όσον αφορά το θέμα των ΡΟΜ και που θέλει να το μελετήσουμε με το σωστότερο τρόπο εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι δύο επιτροπές λοιπόν βρίσκονται σήμερα σε μια διαδικασία η οποία είναι συνεργασίας. Έχουμε την Επιτροπή King Kun στην Επιτροπή Απασχόλησης, η οποία είναι ειδική θα λέμε πάνω σε αυτό το θέμα και η συμβολή της είναι σημαντική. Επίσης, από την Επιτροπή Απασχόλησης, εμείς κάναμε μια ακρόαση με τον Επίτροπο Λάσλο. Από τότε έδειξε ο κύριος Επίτροπος την αποφασιστικότητά του, ούτω ώστε το θέμα των Ρώμα, το θέμα των μη διακρίσεων για τον αγώνα κατά της ε, φτώχειας, για την οποία φτώχεια είναι θύματα αυτή, και προχωράμε περισσότερο από ό,τι είχε γίνει μέχρι τώρα. Από τη δική μας επιτροπή θα έλεγα και το ξέρετε κυρία Επίτροπε ότι για μας δεν είναι, δεν είναι θέμα ενό χαρτιού αυτό, για, να το πώς παράσουμε στην εφαρμογή της στρατηγικής για το 2020 όσον αφορά τον αγώνα κατά της φτώχειας και στον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε τους Ρώμα. Δεν κάνουμε διάκριση. Καμιά φορά κανείς έχει την εντύπωση ότι, ότι σε σχέση με τις κρίσεις που έχουμε θα ξεχαστεί το θέμα, όχι κάθε άλλο. Το πλαίσιο στο οποίο βρισκόμαστε, το κοινωνικό-οικονομικό πλαίσιο εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, ε, έχει να κάνει και με το, θέμα, για το, με το πώς θα λύσουμε το θέμα των Ρώμα. Είναι, έχει συμβολικό χαρακτήρα. Ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε τη φτώχεια και την ένταξη των Ρώμα θα δείξει το στίγμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. την αποφασιστικότητα να αντιμετωπίσει κανεί την φτώχεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εμεί στι δύο, επιτροπέ επιτροπές ε, θα κοιτάξουμε να ορίσουμε το χρονοδιάγραμμα για να μπορέσουμε να πετύχουμε τα μέγιστα και θα το αντιμετωπίσουμε ε, θα συνεχίσουμε μετά από αυτή την ακρόαση τη σημερινή, η οποία είναι ανοιχτή και θετική. Και είναι σημαντική για τα μέλη των δύο επιτροπών μας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Uh, Ευχαριστώ κυρία Μπέρες. Θα ζητήσω καταρχήν από την κυρία Γιάροκα, η οποία ενισχύεται για την έκθεση για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την συμπερίληψη στο Ρωμά, να δώσει την άποψή της και μπορεί φυσικά να αντιδράσει μετά η κυρία Επίτροπος, κυρία Γιάροκα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία αυτή να σας μιλήσω σήμερα. Θα σας παρουσιάσω σύντομα τα πιο βασικά στοιχεία της εκθεσής μου, ώστε να μπορέσουν να έχουν περισσότερο χρόνο ομιλίες και εμπειρογνώμονες και οι εκπρόσωποι των κρατών μελών και της Κομισιόν ε, που θα ε, κάνουν σημαντικές συνεισφορές ε, στη συζήτηση τις επόμενες ε, δύο μέρες. Σημαντικός αριθμός των Ευρωπαίων Ρώμα αντιμετωπίζουν συνθήκες που είναι σχεδόν τελείως απομονωμένες ε, από την γενική οικονομία. Η ε, κοινωνική ένταξη δεν ε, μπορεί να εξεταστεί στα πλαίσια της γενικής πολιτικής. Θα πρέπει να εξετάσουμε τα τεράστια κενά όσον αφορά την, τον σεβασμό των ανθρωπίνων και θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρώπη. Γι' αυτό η στρατηγική των Ρωμά θα πρέπει να βασίζεται στην ε, προώθηση ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεύτερης ε, και τρίτης γενιάς το δικαίωμα απασχόλησης, στέγασης και εκπαίδευσης απαιτεί εξίσου μεγάλη έμφαση με την πρώτη γενιά ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε εξίσου ισχυρή νομική βάση. η, τα περισσότερα έγγραφα που έχουν να κάνουν με τους, Ρώμου, με τους Ρώμα αποτελούν μη ε, δεσμευτικές ε, νομικές προτάσεις. Ε, υπάρχουν κάποιες εθνικές πρωτοβουλίες και καλές προτάσεις τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν ήταν επιτυχής. Το αποτέλεσμα είναι μάλλον αφισβητήσιμο και δείχνει ότι τα μη δεσμευτικά μέτρα ε, δεν αρκούν για την ε, ένταξη των ε, Ρώμα. Χωρίς ισχυρή νομική βάση, χρηματοδοτική υποστήριξη και κίνητρα δεν θα πραγματοποιήσουμε ποτέ τους στόχους μας. Χρειάζεται συντονισμός των δράσεων των ενδιαφερομένων από τις τοπικές κυβερνήσεις μέχρι τα επίπεδα πολλαπλής διακυβέρνησης τα μέσα που ε, αναφέρει η συνθήκη και ο χάρτης ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Θα πρέπει η ευρωπαϊκή στρατηγική το, για τους Ρώμα να υλοποιηθεί. Θα πρέπει να εξετάσουμε την ε, κοινωνική και οικονομική στέρηση των ε, Ρώμα. Η ένταξη μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο αν ε, αντιμετωπίσουμε την ομάδα στόχο της στρατηγικής όχι μόνο με, με βάση τα έθνωτικα χαρακτηριστικά αλλά και τα οικονομικά. Με κανέναν τρόπο δεν ε, θα πρέπει να δημιουργηθούν ε, ε, διαχωρισμοί ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Κατά τη γνώμη μου, δεν χρειάζεται να δημιουργήσουμε κατακαιρματισμένη στρατηγική. Η εποπτεία και η παρακολούθηση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από την Κομισιόν και γι' αυτό, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να διατηρηθεί η ομάδα κρούσης για τους Ρώμα ως, μόνιμη, ως μόνιμος φορέας. Η Κομισιόν θα πρέπει να εξετάζει τα αποτελέσματα των μελτών όταν υποβάλλει προτάσεις προς το Συμβούλιο και ο πίνακας αποτελεσμάτων, το scoreboard δηλαδή ε, για τους Ρώμα θα μπορούσε να αναπτυχθεί. Κάτι ανάλογο με τον πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς. για την υλοποίηση των στόχων της ε, στρατηγικής ε, και για να και ε, με συμβουλευτικό χαρακτήρα προς την ε, Κομισιόν ε, θα πρέπει η Κομισιόν να αναλάβει δράση και πιστεύω ότι έτσι θα μπορούμε να έχουμε και πρακτικά αποτελέσματα. Η φτώχεια και, ο κοινωνικό αποκλεισμό είναι θέματα που βλέπουμε σε όλα τα κράτη-μέλη και ιδιαίτερα σε κάποιες μικροπεριφέρειες. Χρειάζονται λοιπόν ε, αξιόπιστοι δείκτες ώστε να μπορούμε να παρουσιάσουμε ε, την ε, αναλυτική εξέταση της πρόοδου που σημειώνεται. Οι δείκτες αυτοί θα είναι συμπληρωματικά στοιχεία για να αξιολογήσουμε την πρόοδό μας. Κατά τη γνώμη μου χρειάζεται μια ευρωπαϊκή οπτική θα πρέπει να εξετάσουμε την ε, πρόσβαση στην απασχόληση, την ε, σωστή υποδομή, ε, την πρόσβαση στα αστικά κέντρα. Θα πρέπει επίσης να διατεθεί χρηματοδότηση στο επόμενο πολιετές πλαίσιο, ώστε να υπάρχουν πόροι και κίνητρα για την υλοποίηση των μέτρων αποδίδοντας ε, πόρους ε, στα πιο ε, στους πιο κατάλληλους φορείς για την υλοποίηση της στρατηγικής των Ρώμα. Έτσι μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε το αποτέλεσμα. Ο Επίτροπος Χάν έχει αναφερθεί στο θέμα αυτό. Από την άλλη θα υπάρχει σε σύνδεση ανάμεσα στην ε, χρηματοδότηση και στα αποτελέσματα. Αυτές είναι οι βασικές προτεραιότητες που πιστεύω ότι πρέπει να έχει η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τους Ρώμα. Ωστόσο γνωρίζω ότι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική δεν θα αρκεί. Ε, τα λόγια δεν είναι τίποτα χωρίς ε, τις αντίστοιχες ενέργειες και θα πρέπει και οι κυβερνήσεις εκτός των Βρυξελών να ε, κάνουμε κάτι για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Και η συζήτηση αυτή δεν έχει να κάνει μόνο με την ε, στρατηγική για τους Ρώμα, έχει να κάνει και με την ε, αμοιβαία εμπιστοσύνη και την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι ευγνώμων προς τους και όδης που έχουν συμβάλει στην εκπόνηση του κειμένου. Έχουμε πολλές τροπολογίες. Πιστεύουμε ότι η έκθεση αυτή θα είναι ισχυρό μήνυμα προς την Κομισιόν και στο Συμβούλιο σχετικά με το πώς μπορούν να ε, λυθούν τα προβλήματα που θα ε, συζητήσουμε σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Livia. Uh, well, before... Ευχαριστώ πολύ, Λίβια. Πρωτού το δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Επίτροπη. Θα παρακαλέσω να κάνετε λίγη ησυχία. Είναι πολύ δύσκολο να εργάζεται κανείς σε αυτήν την αίθουσα με τη συνεχή βαβούρα η οποία επικρατεί μερικέ φορέ. Η Αντιπρόεδρος τη Επιτροπή η κυρία Ρέτινγκ, έχει το λόγο τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ εξ αρχή να σας πω πόσο ευγνώμων είμαι που τροποποίησατε την ημέρησια διάταξη για να έχω τη δυνατότητα να μιλήσω. Δεν έκανα αυτό που μου είπε ο γιατρός μου, που μου είπε να μείνω στο κρεβάτι μου. Θεώρησα ότι ήταν σημαντικό να έρθω εδώ, παρά το γεγονό ότι δεν μπορώ να μείνω πολλή ώρα. Παρακαλώ να κατανοήσετε το προσωπικό μου είναι εδώ, οι υπηρεσίε μου θα καταγράψουν όλα αυτά τα οποία θα πείτε. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων που και πάλι γίνεται αυτή η συνεδρίαση από κοινού από την Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών και την Επιτροπή Απασχόληση κάθε νόημα έχει αυτό και επίση χαίρομαι ιδιαίτερα για την παρουσίαση της Λίβια Ζαρόκα ως εισηγήτρια. Υπάρχουν πολλά στοιχεία στην παρουσίαση της εισηγήτριας που θα δώσω στο, στους συναδέλφους, στον κύριο Άντορ και στον κύριο Χάν που είναι αρμόδια επιτροπή σε άλλα θέματα, το θέμα των μικροπεριφερειών και τον αποκλεισμό εκεί και επίση τη σύνδεση μεταξύ μικροχρηματοδότηση και αποτελεσμάτων. Μια ανάλυση λοιπόν εκ των υστέρων και όχι μόνο μια ανάλυση εκ των προτέρων όπως κάνουμε. Αυτό επομένως είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο εάν ο κύριος Άντορ και ο κύριος Χάν εξετάσουν τους κανόνες που διέπουν το Κοινωνικό και Περιφερειακό Ταμείο. Η πρόταση τώρα για την οποία η κυρία Γιαρόκα είναι εισηγήτρια αναφέρεται άμεσα σε μένα γιατί δεν αφορά τη δημιουργία ενός μόνιμου φορέα αλλά για να αναλάβει η ομάδα κρούσης για τους Ρώμα την ευθύνη να συνεχίσει να δει τι γίνεται στις περιφέρειες της Ευρώπης, τι γίνεται σε επίπεδο βάσης, να μπορέσει να έρθει σε επαφή με τα εθνικά σημεία επαφής για να μπορεί να ανταλλάσσει απόψεις και να συλλέγει πληροφορίες. Αυτό μου φαίνεται μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση και είναι κάτι το οποίο θα αναλύσω και έχω ήδη μια πάρα πολύ θετική άποψη για αυτή την πρότασή σας. Και αγαπητά μέλη των δύο κοινοβουλευτικών επιτροπών, ξέρετε ότι και από την αρχή της θητείας μου, εγώ έχω συνεργαστεί στενά μαζί σας για να εξασφαλίσουμε ότι η συμπερίληψη των Ρωμά στην κοινωνία μας, η οποία έχει τεθεί στην ημερησία διάταξη, αλλά δεν έχει αντιμετωπιστεί στην πράξη από τα περισσότερα κράτη-μέλη, θέλω να αναβαθμιστεί αυτή η στρατηγική συμπερίληψη. Έχουμε πολλά πράγματα να πράξουμε και ξέρω ότι αυτή η εργασία δεν μπορεί να περατωθεί σε τρεις εβδομάδες. Θα χρειαστούμε χρόνια για να μπορέσουμε να δρέψουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Και έτσι βλέπω και με μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι η Επιτροπή Πολιτισμού η οποία καλύπτει και τα θέματα παιδείας, ότι εξετάζει το ζήτημα της προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης. Νομίζω λοιπόν ότι αυτά είναι εξόχως σημαντικά στοιχεία για να μην χάσουμε την επόμενη γενιά των ε, Ρωμά στην Ευρώπη Πρέπει επομένω να εστιάσουμε την προσοχή μας σε όλα αυτά τα ζητήματα. Ξέρουμε ότι το να ξεπεραστούν δεκαετίες κοινωνικού αποκλεισμού είναι κάτι που θα απαιτήσει μεγάλη αποφασιστικότητα και χαίρομαι που έχω το Κοινοβούλιο μαζί μου στον αγώνα αυτό. Όπως είπε όμως σωστά και η συγγήτρη, αυτό το οποίο λείπει δεν είναι άλλο ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για να λύσουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι σε επίπεδο βάσης να εργαστούμε σκληρά εκεί που βρίσκεται το πρόβλημα. Στις μικρο περιφέρειες όπως λέει η Λίβια, εκεί είναι που πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Και είμαι ευγνώμων όπως είπα και προηγουμένως προς τη Βελική Προεδρία η οποία έχει δημιουργήσει μια πλατφόρμα για τους Ρωμά και την έχει εσωματώσει στην ημερησία διαταξή τη και προστοκώ στην επερχόμενη Ουγγρική Προεδρία και εξάλλου ο υπουργό ο οποίος είναι αρμόδιος για τα θέματα αυτά είναι μαζί μας σήμερα και είναι μια ευκαιρία να έρθει και πάλι το θέμα αυτό στην ημερησία διαταξή. Επομένως, στους επόμενους μήνες δεν θα έχουμε μόνο μία ή δύο επιτροπές που θα εξετάζουν το θέμα αυτό, αλλά ένα σύνολο φορέων που θα αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα, όχι μόνο η Κοινωνική Επιτροπή, η Επιτροπή Δημοσίου Ελευθεριών, η Επιτροπή Παιδείας, Εκπαίδευσης και Κουλτούρας και διάφοροι σχηματισμοί του Συμβουλίου θα αντιμετωπίσουν υπό το δικό του πρίσμα το, ο κάθε σχηματισμός το πρόβλημα αυτό. Και αυτό είναι ένα σημαντικό καινοτόμο βήμα. Ποτέ δεν είχε ξαναγίνει κάτι τέτοιο στο παρελθόν και όλα αυτά μπορούν φυσικά να αυξήσουν την αποτελεσματικότητά μας στην πράξη. Στην πράξη σημαίνει στις χώρες προέλευσης, στις χώρες υποδοχής, σε εθνικό, σε περιφερειακό, σε τοπικό επίπεδο. Τον τελευταίο καιρό στην Κομισιόν έχουμε κάνει μεγάλες προσπάθειες να αναπτύξουμε καινοτόμους μηχανισμούς για να βρούμε και τρόπους να δώσουμε υποστήριξη στα κράτη-μέλη για την καλύτερη συμπερίληψη και ενσωμάτωση στην κοινωνία των Ρωμά, Θυμόσαστε όλη την ανακοίνωση της Κομισιόν για την Κοινωνική και Οικονομική Ενσωμάτωση που εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2010, που θεσπίζει μια σειρά από προτεραιότητες για δράση. Ξέρετε επίσης τι έχει γίνει μεταξύ του Απριλίου και αυτής της στιγμής. Δεν χρειάζεται να επανέλθουμε, αλλά είναι γεγονός ότι η ομάδα κρούσης για τους Ρωμά που ξεκίνησε τις εργασίες της το Σεπτέμβριο του έτους συνεδριάζει τακτικά για να μπορέσει να εξετάσει την αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης και των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως την κατεύθυνση της ενσωμάτωσης των Ρωμά. Θέλω να κάνω μια προσωπική παρατήρηση και αναφέρομαι κατευθείαν στα μέλη της Επιτροπής, των Επιτροπών αυτών που έρχονται από διάφορα κράτη-μέλη. Θα έχει μεγάλη δυσκολία η Κομισιόν να σας δώσει σημαντικά και θετικά αποτελέσματα αν όλα τα κράτη-μέλη δεν μας βοηθήσουν με το να μας παράσχουν τις απαραίτητες πληροφορίες. Κάνω μια έκκληση λοιπόν σε όλους τους κοινοβουλευτικούς που είναι εδώ, όχι μονάχα να ορθώσουν το ανάστημά τους και τη φωνή τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και στην ίδια τη χώρα τους να υπεθυμίσουν στις κυβερνήσεις τους ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία σε αυτό το εγχείρημα. τη βάση λοιπόν του έργου της ομάδας κρούσεως για τους Ρώμα, θα παρουσιάσουμε τον, την Άνοιξη ένα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για, την, για τις εθνικές στρατηγικές ενσωμάτωσης των Ρωμά. Η κάθε λέξη μετράει. Γιατί άκουσα προσεκτικά αυτά που είπε η συγγητριά σα. Δεν αρκεί να έχει κάνει ένα πλαίσιο που δεν έχει τίποτα μέσα. Γι' αυτό λέω ένα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης ή ενσωμάτωσης των Ρωμά. Η δουλειά θα πρέπει να γίνει εκεί που βρίσκεται το πρόβλημα και θέλω να τονίσω ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τις χώρες από τις οποίες προέρχονται οι Ρωμά, αλλά και στις χώρες υποδοχής. Περιλαμβάνω λοιπόν μέσα στην στρατηγική αυτή 27 κράτη-μέλη. Γνωρίζουν φυσικά ότι το πρόβλημα στην πατρίδα μου το Λουξεμβούργο είναι λιγότερο σημαντικό από ό,τι είναι στις δικές σας χώρες και ιδίως στην ε, χώρα της προέλευσης της εισηγήτριας, στην Ουγγαρία. Αλλά η κάθε χώρα θα πρέπει να επιλύσει τα δικά της προβλήματα. Αυτό λοιπόν το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Εθνικές Στρατηγικές Ενσωμάτωσης στο Ρώμα θα παρουσιαστεί τον Απρίλιο του 2011. Και έτσι θα είναι έτοιμο για την πλατφόρμα των Ρωμά. Νομίζω ότι θα γίνει αυτό 8 Απριλίου, αν θυμάμαι καλά. Θα έχουμε λοιπόν αυτή τη στρατηγική έτοιμη για του χρόνου, ώστε όχι μόνο να συζητηθούν αυτά στην πλατφόρμα για τους Ρωμά, αλλά για να πάμε στους διάφορους σχηματισμούς του Συμβουλίου, όπως είπα προηγουμένως, και βασίζομαι εδώ στη συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για να, παρίσταται, να παρίστανται τα μέλη ε, του Κοινοβουλίου στις διάφορες επιτροπές και να εξετάσουν ενδελεχώς το θέμα αυτό. Ξέχουμε, ξέρετε ότι έχουμε στείλει στα μέλη τα ερωτηματολόγια για τη χρήση των εθνικών και ευρωπαϊκών ποσών για την ενσωμάτωση των Ρωμά και η Κομισιόν αυτή τη στιγμή αναλύει προσεκτικά τις απαντήσεις που έχουμε ήδη λάβει από τα κρατη για το θέμα αυτό. Η επόμενη πλατφόρμα για τους Ρωμά θα λάβει χώρα στις 13 Δεκεμβρίου και όπως σας είπα, όπως είπα προηγουμένως και κάνω μια άμεση σύνδεση με αυτά που είπα προηγουμένως. Γιατί αυτή η πλατφόρμα για τους Ρωμά θα αναλύσει ένα από αυτά που εγώ θεωρώ ότι είναι τα βασικά προβλήματα που είναι τα προβλήματα της νεαρής παιδικής ηλικίας πώς τα παιδιά των Ρωμά μπορούν να ενσωματωθούν στα συστήματα παιδείας. Η Ουγγρική Πρεσβεία, συγγνώμη, η Ουγγρική Προεδρία θα συνεχίσει λοιπόν με την επόμενη πλατφόρμα και εξακολουθούμε να οργανώνουμε γεγονότα για αύξηση της συνειδητοποίησης σε σχέση με τη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενσωμάτωση στο Ρωμά. Είχαμε τέτοιες εκδηλώσεις στη Ρουμανία, θα έχουμε και στη Σλοβακία και τη Βουλγαρία. Αλλά και πάλι αντιδρώντας αυτά που είπε η συγγήτριά σας, πρέπει να πω ότι δεν μπορούμε να δούμε το θέμα μονάχα από την οπτική γωνία της χρηματοδότησης. Όταν αντιμετωπίζουμε το ζήτημα των Ρωμά πρέπει να δούμε και το θέμα και από το πρίσμα, υπό το πρίσμα των δικαιωμάτων τους και να εξασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματα που περιλαμβάνει η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πράγματι εφαρμόζονται και σε εθνικό επίπεδο. Αν δεν υπάρχει λοιπόν μια ισότηση μεταξύ όλων των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορούν να εφαρμοστούν αυτά τα δικαιώματα και οι Ρωμανοί και αυτοί οι Ευρωπαίοι πολίτες. Και έρχομαι τώρα στο θέμα της Γαλλίας για να προλάβω, να αποκαταλάβω ένα ερώτημα το οποίο σίγουρα θα μου θέσετε. Θυμόσαστε πολύ καλά ότι ζητήσαμε από τις γαλλικές αρχές να μεταφέρουν ε, διαδικαστικές εγγυήσεις και νομικές προδιαγραφές, όπως αναφέρονται στην Οδηγία 2004 για την ελεύθερη κυκλοφορία, στη γαλλική νομοθεσία, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζονται με έναν τρόπο ο οποίος είναι δίκαιος, αναλογικός και μη διακριτικός τρόπος και πάνω απ' όλα όταν αυτοί εμπλέκονται σε καταστάσεις συγκρουσιακού χαρακτήρα. Είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ασφάλεια δικαίου που προνοεί η οδηγία του 2004. Νομικές και διαδικαστικές διασφαλίσεις. Μετά από την παρέμβαση της Κομισιόν, 15 Οκτωβρίου, 15 Οκτωβρίου, η γαλλική κυβέρνηση μας έδωσε λεπτομερή τεκμηρίωση η οποία περιλαμβάνει και ένα σχέδιο νόμου και άλλα μέτρα και ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για να εφαρμοστούν αυτές οι εγγυήσεις και διασφαλίσεις βάσει της οδηγίας του 2004 να μπουν στη γαλλική νομοθεσία μέχρι τις αρχές του 2011. Η Γαλλία λοιπόν έκανε ακριβώς ό,τι της είχε ζητήσει η Κομισιόν και υπευσικά ότι θα το πράξει αυτό και εμείς μέχρι τότε θα παρακολουθούμε τον τρόπο μεταγραφής της οδηγίας για την ελεύθερη κυκλοφορία και συγχρόνως παρακολουθούμε και την εφαρμογή των βασικών κανόνων που περιέχονται σε αυτήν την οδηγία, όχι μόνο στη Γαλλία, αλλά και σε όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορώ ήδη να σας πω ότι ξεκίνησα συζητήσεις με περίπου 20 κράτη-μέλη σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο η οδηγία για την ελεύθερη κυκλοφορία έχει εφαρμοστεί ή κάποιες φορές δεν έχει εφαρμοστεί και μπορώ να σας πληροφορήσω ότι τα κράτη-μέλη κινούνται με μεγάλη ταχύτητα για να επιλύσουν τα εκκρεμούντα ακόμα προβλήματα της ε, εφαρμογής αυτής της οδηγίας. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της οδηγίας αυτής και την, ε, μεταγραφή της στο εθνικό δίκαιο. Το άλλο πρόβλημα είναι η εφαρμογή της οδηγίας, της οδηγίας αυτής στην πράξη. Και εδώ οι γαλλικές ε, αρχές μας έδωσαν λεπτομεριακά στοιχεία για τη δράση των γαλλικών αρχών σε σχέση με τα γεγονότα φέτος το καλοκαίρι. Έχουν αναλύσει αυτό το υλικό υπηρεσίες Κομισιόν και καταλήξαμε στο εξή συμπέρασμα. Η εξέταση των ε, ατομικών καταστάσεων των εμπλεκομένων ατόμων δεν φαίνεται να έχει γίνει με συστηματικό τρόπο. Ιδίω όταν εκδίδονται εντολές αποχώρησης από το γαλλικό έδαφος λόγω έλλειψης επαρκών πόρων. Δεύτερον, η ατομική αξιολόγηση της απειλής που αποτελούν τα άτομα αυτά για τη δημόσια τάξη στο φως προηγούμενων ε, ποινικών υποθέσεων και καταδικών δεν έγιναν στο φως της οδηγίας και των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου. Η ανακοινωθήσα μεταγραφή από τη Γαλλία των προνοιών περί διαδικαστικών και ουσιαστικών σε νομικό επίπεδο διασφαλίσεων Κατά την άποψη των εμπειρογνώμων της Κομισιόν θα πρέπει να δώσουν τέρμα σε αυτές τις ενέργειες της γαλλικής, των γαλλικών αρχών στο μέλλον. Και γι' αυτό απαιτεί ε, η Κομισιόν μέχρι την άνοιξη του 2011 να εφαρμοστεί, να μεταγραφεί πλήρω η οδηγία του 2004, όπω συμφωνήθηκε και από τη Γαλλία, γιατί αυτό αποτελεί την καλύτερη εξασφάλιση και για το μέλλον. Να υπογραμμίσω για μια ακόμα φορά ενώπιον των κοινοβουλευτικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενώπιον του Βέλγου, ενώπιον της Βελγίδος Υπουργού, εδώ είναι, και τον Υφυπουργό, τον αρμόδιο το Βέλγο, θέλω να τονίσω και πάλι ότι θέλουμε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τη δέσμευσή μας για την επίλυση αυτών των προβλημάτων και ο στόχος μας είναι να μπορούμε να πούμε σε μερικά χρόνια ότι επήλθε σημαντική πρόοδος σε απτούς όρους για τα θέματα αυτά. Στους τομείς δηλαδή όπου το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει. Φυσικά μας ενδιαφέρει για το πώς η μεγαλύτερη μειονότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση την χάνει αντιμετώπιση από τα κράτη-μέλη και πώς μπορεί να εξέλθει από την παγίδα ένδυας μέσα στην οποία υπάρχει ένα μεγάλο μέρος αυτής της μειονότητας πώς πρέπει να εξέλθουν από αυτή την παγίδα ένδυας. Μαζί με τον συνάδελφό μου λοιπόν τον κύριο Λάσλο Άντορ, ο οποίος είναι ο αρμόδιος για την Ευρώπη 2020, τη στρατηγική αυτή, η οποία συμπεριλαμβάνει και τον αγώνα κατά της ένδυας, ο οποίος είναι πολύ σημαντικό στοιχείο αυτής της πολιτικής. Ο στόχος μας είναι να εργαστούμε για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τους κανόνες δράσης που ελπίζουμε ότι στη συνέχεια θα εφαρμοστούν και στην πράξη από τις κυβερνήσεις και τις περιφέρειες με μεγάλη ταχύτητα. Η πίεση λοιπόν που ασκείται από το Κοινοβούλιο και από τα διάφορα από τις διάφορους σχηματισμούς του Συμβουλίου είναι πάρα πολύ μεγάλη για να μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτό το στόχο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. And thank you that you didn't listen to your uh, doctor. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεν ακούσατε το γιατρό σας. Τώρα να επανέλθουμε στην ε, κανονική σειρά των ομιλητών. Καταρχήν να ζητήσω από την κυρία Κίνγκα Κόνς να παρέμβει. Είναι η, η συντάκτρια της νομοδότησης ε, για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική ε, για την ένταξη των Ρώμα ε, στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ πολύ. Βρίσκομαι εδώ, όπως είπατε, με δύο διαφορετικές ε, ιδιότητες. Είμαι η συντάκτρια της γνωμοδότησης, ε, αλλά είμαι και σκιώδης εισηγήτρια στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Θα ήθελα λοιπόν να πω λίγα λόγια και για τις δύο πτυχές του προγράμματος αυτού που συζητάμε. Στην αρχή αναφέρθηκε ότι πολλά έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες. Δεν θα ήθελα να επαναλάβω όλο τον κατάλογο. Να πω ότι από πλευράς του Κοινοβουλίου σημαντικό ήταν το ψήφισμα μετά την απέλαση των Ρώμα από τη Γαλλία. Και τώρα ακούσαμε ότι έγιναν και άλλα βήματα έκτοτε. Το Κοινοβούλιο ε, θεώρησε ότι ε, ε, έτσι παραβιάζονταν θεμελιώδη δικαιώματα και ανθρώπινα δικαιώματα. Όσον αφορά την έκθεση αυτή, να μιλήσω και με τις δύο μου όπως είπα. όσον αφορά το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το θέμα καταπολέμησης των διακρίσεων. Θα πρέπει να πούμε σαφώς ότι η Ρώμα είναι Ευρωπαίοι πολίτες με ίσα δικαιώματα. Δεν είναι λοιπόν αποδεκτή καμία διάκριση ούτε στα κράτη-μέλη ούτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γνωρίζουμε ότι γίνονται πολλές διακρίσεις όσον αφορά τη στέγαση, όσον αφορά την εκπαίδευση. Είμαι σίγουρη ότι η έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού ε, αναφέρει αυτό και σε άλλα επίπεδα και όσον αφορά δηλαδή το δικαίωμα της ε, ελεύθερης κινητικότητας. Θα χρειαστούμε λοιπόν Έχουμε λοιπόν ε, την ε, οδηγία για την καταπολέμηση των διακρίσεων, η οποία είναι οριζόντια. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Το επόμενο ε, θέμα θα είναι η υλοποίηση της οδηγίας. Όσον αφορά τις κοινωνικο-οικονομικές πτυχές, όλοι γνωρίζουμε ότι στην έκθεση αυτή αναζητούμε τρόπους να πετύχουμε το στόχο μας. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολύ καλές πρωτοβουλίες, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποιοι διαθέσιμοι πόροι, δεν αρκούν όμως για να φτάσουμε τους ανθρώπους ε, που ε, υποφέρουν περισσότερα, που ε, ζουν απομονωμένοι κλπ. Στη στρατηγική 2020, λοιπόν, 2020, σε επίπεδο κρατών μελών, ε, όσον αφορά το κεφάλαιο της ένταξης, θα πρέπει να, ε, της κοινωνικής ολοκλήρωσης, θα πρέπει να αναφέρουμε και την, ένταξη, την κοινωνική ένταξη των Ρώμα. Θα πρέπει να παρακολουθούμε τα αποτελέσματα, τον αντίκτυπο, ε, διότι συχνά δεν εξετάζουμε το πραγματικό αντίκτυπο των μέτρων που λαμβάνουμε. Πιστεύω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε βήμα-βήμα, με μια πρόσβαση όχι βασισμένη σε προγράμματα, αλλά να έχουμε πολύπλοκα ε, προγράμματα τα οποία να λαμβάνει υπόψη την απασχόληση, τη στέγαση, την εκπαίδευση, διότι αν θέλουμε να πετύχουμε πρόοδο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όλα τα στοιχεία αυτά. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πολύ σημαντικό να ληφθούν αποφάσεις ε, σχετικά με τους ε, πόρους. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, την πτυχή των διακρίσεων. Εάν δεν έχουμε το στοιχείο της αιρεσιμότητας, δεν θα φτάσουν ποτέ οι πόροι αυτοί στις κοινότητες των Ρώμα. Αναφέρθηκα στη στενή παρακολούθηση που θα βασίζεται σε μελέτες αντικτύπου. Χρειαζόμαστε ανεξάρτητους ε, ε, ε, παρατηρητές και χρειαζόμαστε όρους αναφοράς που θα αποτελέσουν τη βάση της παρακολούθησης αυτής. Για να πετύχουμε πρόοδο όμως σε κάποια χρόνια χρειαζόμαστε μία κοινή εγκάρσια και συντονισμένη προσπάθεια ώστε να μπορέσουμε να ε, έρθουμε σε επαφή με ε, αρχές σε τοπικό επίπεδο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να πετύχουμε τη συμμετοχή των ε, Ρώμα και να αυξηθεί η αφοσίωση για την επίλυση του θέματος στα διάφορα επίπεδα. Θα ήθελα να αναφερθώ στις ε, ε, πρόοδους που έχει που έχουν σημειωθεί. Έχουμε την έκθεση της ε, Υπηρεσίας για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Έχουμε αρχίσει να επισκεφτόμαστε τις χώρες ε, τον Ρώμα, να τους δούμε από κοντά, να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα. Υπάρχουν όμως και διεθνείς οργανισμοί, ο ΣΑ, το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, που παρακολουθούν τι πραγματικά συμβαίνει στις διάφορες χώρες. Χρειαζόμαστε συνεχιζόμενη ανάδραση όσον αφορά του, τα αποτελέσματα, τα επιτεύγματα για να μπορούμε να βλέπουμε σωστά αποτελέσματα. Και θα ήθελα να καλέσω όσους βρίσκονται εδώ στην αίθουσα ε, να βοηθήσουν στη διαδικασία αυτή και να συνεργαστούμε στενά για την επίλυση των θεμάτων αυτών. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Mrs. Ευχαριστώ κύριε Γκέντς. Δύο ακόμα συνάδελφοι <clears throat> θα λάβουν το λόγο. Ο κύριος Χάνου Τακκουλά ο οποίος είναι ο συντάξης γνωμοδότησης στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας και ο κύριος Κόβατσεφ, ο οποίος είναι ο συντάκτης γνωμοδότησης στην Επιτροπή Περιφερειακών Θεμάτων. Μετά από τους δύο συναδέλφους θα δώσω το λόγο στους εκπροσώπους της Βελγικής και της επερχόμενης Ουγγρικής Προεδρίας και μετά θα αρχίσει η ανταλλαγή ερωτήσεων και απαντήσεων. Υπάρχει ίσως μια παρεξήγηση μεταξύ σας για το πώς θα γίνει κάτι τέτοιο και ποια ήταν η σειρά του προγράμματος, αλλά η προτεραιότητα θα δοθεί στους ε, συναδέλφους που είναι αρμόδιοι γνωμοδοτήσεων στις διάφορες ε, επιτροπές, μετά η Προεδρία και μετά ακολουθούν οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις. Έχετε το λόγο κύριε Τάκουλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Χαίρομαι που είμαι εδώ σήμερα, στο τόσο σημαντικό αυτό σεμινάριο και θέλω να, ευχαριστήσω τους οργανωτές αυτού του σεμιναρίου για την οργάνωση αυτή και για το γεγονός ότι μου έδωσαν και τη δυνατότητα να λάβω το λόγο. Για πολύ καιρό νομίζω ότι αυτό το θέμα το είχαμε καταχωνιάσει κατά το χαλί, γιατί δεν είναι από τα ευκολότερα προβλήματα να επιλύσει κανείς. Γνωρίζω πολύ καλά την πολυπλοκότητα του θέματος αυτού για την Κομισιόν και για τα κράτη-μέλη και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την ανάγκη να έχουμε μια ολιστική αντιμετώπιση. Δεν μπορούμε να θέσουμε όλα τα αυγά στο ίδιο καλάθι. Επειδή έχω λίγα λεφτά μονάχα θα εστιάσω την παρέμβασή μου στις εκπαιδευτικές πτυχές του προβλήματος αυτού. Επειδή είμαι και ο εισηγητής της Επιτροπής Πολιτισμού για τη στρατηγική συμπερίληψη των Ρωμά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τελευταίο χρόνο εγώ ενεπλάκην και σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ε, παιδιών Ρωμά στο Βουκουρέστι, στη Ρουμανία, που προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τις βέλτιστες πρακτικές από τη Φιλανδία στο πρόγραμμα σπουδών. Δεν έχω στόχο το να υποτιμήσω άλλες περιοχές δράσης. Πιστεύω όμως ότι η παιδεία είναι από τα πιο σημαντικά θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε όταν μιλάμε για τη συμπερίληψη των Ρώμα. Οι περισσότεροι θα συμφωνούσαν ότι για ένα άτομο η παιδεία είναι ο κύριος συντελεστής, συντελεστής της μελλοντική του προόδου και επιτυχίας. Θα πρέπει λοιπόν τα πρότυπα της εκπαίδευσης να είναι ε, ως τον ετών πιο υψηλά και να μην αντιμετωπίσουν τα παιδιά των Ρωμά διακρίσεις. Πρέπει λοιπόν να δοθούν ιδιαίτερα κονδύλια στην, ε, να δοθούν, να δοθούν επενδύσεις στην εκπαίδευση των παιδιών Ρωμά. Θα πρέπει οι αρχές να κάνουν προσπάθειες να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή των παιδιών <clears throat> το Ρωμά στην ευρωπαϊκή παιδεία και ιδίως το ότι θα μείνουν στο σχολείο μέχρι την ηλικία που είναι υποχρεωτική εκπαίδευση. Υπάρχει υψηλός βαθμός απουσιών των παιδιών Ρωμά Εν μέρει γιατί οι γονείς δεν κατανοούν τη σημασία της παιδείας, αλλά υπάρχουν και άλλα προβλήματα όπως είναι η ένδια, ο διαχωρισμός, οι διακρίσεις. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να εμπλέξουμε καλύτερα τους γονείς και αυτούς στον διάλογο αυτό. Υπάρχει πίεση στις κοπέλες και τις γυναίκες Ρωμά να φύγουν από το σχολείο και είναι απαραίτητο να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα για να εξασφαλίσουμε ότι είναι σωστά εκπαιδευμένοι οι διδάσκοντες ώστε να κατανοήσουν πώς λειτουργούν τα παιδιά των Ρωμά και οι γονείς τους. Είναι σημαντικό να έχουμε λοιπόν και μία μεταλαμπάδευση βελτίστων πρακτικών. Έχουμε μιλήσει για το θέμα αυτό στην ε, εκπαίδευση, αλλά στην πράξη γίνονται πολύ λίγα πράγματα στον τομέα αυτό. Θα μπορούσα να πω πολύ περισσότερα, απλώ όμω θέλω να κλείσω τονίζοντα και το πόσο πλούσιε είναι οι πολιτιστικέ παραδόσει των Ρωμά. Αν είμαστε πραγματικά ειλικρινεί, θα πρέπει να παραδεχτούμε όλοι ότι ξέρουμε ελάχιστα πράγματα για το ποιοι είναι οι Ρωμά, τα 10 εκατομμύρια Ρωμά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να παροτρύνουμε τον κόσμο να έχει μια καλύτερη κατανόηση αυτού του πολιτισμού μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κουλτούρα και ο πολιτισμός δεν πρέπει να τεθούν στο περιθώριο όταν συζητούμε τη συμπερίληψη των Ρωμά στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Τάκουλα. Κύριε Κόβατσεφ, είστε το επόμενο ομιλητή. Συντάκτη νομοδότηση στην Περιφερειακή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω που οργανώσατε την ακρόαση αυτή. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο και να μην επαναλάβω αυτά που είπαν οι συνάδελφοι, αλλά να σας παρουσιάσω τις θέσεις που συζητήσαμε στην Επιτροπή Περιφερική Ανάπτυξης. Είμαι εισηγητής της έκθεσης, ε, στην έκθεση αυτή για την Ευρωπαϊκή Στατική για την κοινωνική ένταξη των Ρώμα. Περίπου 12 εκατομμύρια, υπάρχουν διάφορα νούμερα, αλλά ίσως αυτό είναι το ε, σωστό νούμερο. Ζουν στην Ευρώπη, ε, τόσοι Ρώμα ζουν στην Ευρώπη, με πολύ ξεχωριστό τρόπο ζωής. Δυστυχώς, μεγάλος αριθμός της μειονότητας αυτής ε, ζει σε συνθήκες μεγάλης ε, φτώχειας ε, και κοινωνικής και, οικονομικής, και κοινωνικού αποκλεισμού. Δεν μπορεί να υπάρξει μία λύση που να ταιριάζει σε όλου ε, για του ε, Ρώμα, όπω μόλι είπε η Επιτροπό ε, Ρέντινγκ. Πρέπει τοπικά να γίνει δουλειά εκεί που βρίσκονται και τα προβλήματα. Ζούμε όμως στην Ευρώπη, μία Ευρώπη χωρί σύνορα, την Ευρώπη τη ελευθερία και της ευημερία και γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να συντονιστούν τα μέτρα σε ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο για να αντιμετωπίσουμε τις ε, προκλήσεις αυτές. Ας μιλήσουμε καταρχήν για τη στέγαση. Την άνοιξη του 2010 η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ε, διέπρινε τη δυνατότητα στέγασης ε, και για περιθωριοποιημένους ε, κοινότητες, ιδιαίτερα ε, για, την, ε, για τις κοινότητες ε, των Ρώμα. Τα κράτη-μέλη μπορούν να αναθεωρήσουν τα τοπικά τους προγράμματα και να δώσουν νέες προτεραιότητες στις επενδύσεις χρησιμοποιώντας πόρους από, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Δυστυχώς έχουμε μάθει ότι κανένα κράτος μέλος μέχρι τώρα δεν έχει χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα αυτή. Εάν πρέπει να αλλάξουμε κάτι, θα θέλαμε το κράτη μέλη να μα το πούνε αυτό. Εάν η συγχρηματοδότηση αποτελεί πρόβλημα, κάτι που συζητήσαμε σήμερα στην Επιτροπή Περιφερειακή Ανάπτυξη, α ξεκινήσουμε με 100% ε, χρηματοδότηση και όχι συγχρηματοδότηση. Η παρούσα κατάσταση ε, στην ε, στέγαση των Ρώμα δεν είναι καλή, διότι υπάρχουν πόροι, αλλά τα χρήματα αυτά δεν χρησιμοποιούνται για να λυθεί το πρόβλημα. Η γνώμη τη Επιτροπή Περιφερειακή Ανάπτυξη είναι ότι χρειάζεται απλοποίηση στη χρήση των πόρων αυτών. Η χρηματοδότηση για τη στέγαση είναι μια ευκαιρία να συμπληρωθούν οι προσπάθειες ε, των ε, εθνικών αρχών ε, για να επιτευχθεί η κοινωνική ένταξη των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων εντός της Ευρώπης. Μπορούμε να κάνουμε πολλά όσον αφορά την στέγαση των Ρώμα. Μπορούμε να βελτιώσουμε την υποδομή της υπηρεσίας κοινής ωφελίας και άλλα αποτελεσματικότητα των μέτρων ε, έχουμε όταν ε, διδάσκουμε τον κόσμο να ψαρεύει και όχι όταν τους δίνουμε ψάρια. Πιστεύω λοιπόν ότι η χρηματοδότηση της στέγασης θα πρέπει να συνδέεται με κάποιες ε, προϋποθέσεις που να έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση των παιδιών και άλλες. Διότι η κοινωνική ένταξη για μας θα πρέπει να είναι μια αμοιβαία διαδικασία θα πρέπει και οι μειονότητε, ε, αλλά και το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού να επιθυμούν την ε, ένταξη αυτή. Ε, όλα αυτά αποτελούν οικονομική ανάγκη, δεν υπάρχει εναλλακτική λύση στην ένταξη το Ρώμα, όχι για λόγους φιλαθροπίας, αλλά λόγω των ε, συμφερόντων των κρατών μελών. Όλοι οι πολίτες, οι επιχειρήσεις ε, και η κυβέρνηση ε, ωφελούνται από ένα μεγαλύτερο εργατικό δυναμικό. Η ένταξη το Ρώμα αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της Ουγγρικής Προεδρίας και η, Ευρώ... Στρατηγική Ευρώπη 2020 σχετίζεται πολύ με το θέμα αυτό. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το... την πρόορη εγκατάλειψη του σχολείου και άλλα προβλήματα στα πλαίσια της στρατηγικής 2020. Δεν χρειάζεται να επανεφεύγουμε τον τροχό, δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε τα ίδια θέματα, αλλά μέσα στα τελευταία 10 χρόνια ακούσαμε πολλά, πολλά σχέδια δράσης, πολλές στρατηγικές για τους Ρώμα, δυστυχώς όμως με ελάχιστο αποτέλεσμα. Ελπίζουμε λοιπόν ότι τώρα με μια συντονισμένη ε, προσπάθεια από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωσης και των κρατών μελών θα έχουμε ε, πιο καλό αποτέλεσμα. Η οικονομική κρίση έχει αυξήσει τις δυσκολίες που δημιουργεί η φτώχεια, η έλλειψη δεξιοτήτων όμως ε, και εκπαίδευσης που είναι υπεύθυνα για τον είναι υπεύθυνα για, την, για τον κοινωνικό αποκλεισμό. Θα ήθελα να τονίσω ότι υπάρχουν προσπάθειες Ευρωπαϊκής Ένωσης για να καταπολεμηθεί η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός που θα συνεχιστούν και μετά το 2013. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Κοβάτσεφ. Και τώρα στρέφουμε προς το Συμβούλιο. Έχουμε τη, τους εκπροσώπους των, της τωρινής και της επομένης ε, Προεδρίας. Θα ζητήσω καταρχήν από την κυρία Ζουέλ Μιλκέ, που είναι Υπουργός Απασχόλησης και Ίσων Ευκαιριών στο Βέλιο, να μας παρουσιάσει τις απόψεις της και μετά ο κ. Ζόλτιν Μπάλοφ, ο οποίος εκπροσωπεί την επερχόμενη ε, Προεδρία της Ουγγαρίας. Κυρία Μιλκέ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν να ευχαριστήσω για την πρόσκληση εδώ που καλέσατε την ε, δημόσια κρόαση μας καλέσατε σαν φελική ε, προεδρία για το θέμα των Ρώμα Νομίζω ότι θέλουμε να δείξουμε ότι η Ρώμα είναι μια προτεραιότητα στο διάλογο των ευρωπαικων ξερουμε Ξέρουμε ότι 10-12 εκατομμύρια είναι η Ρώμα στην Ευρώπη και η πλειοψηφία αυτών αποτελούν Ευρωπαίους πολίτες, άρα δεν τίθεται το θέμα. Συχνά ζουν κάτω από συνθήκες που είναι ιδιαίτερα ανθρωπές. και επίσης αποτελούν ένα, θα λέγαμε, ευπαθές γκρουπ ε, ανθρώπων, υπάρχει μεγάλη ανεργία, ε, άσχημες συνθήκες ε, ε όχι καλή πρόσβαση στην περίθαλψη. Γι' αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι φυσικά θύματα του κοινωνικού αποκλεισμού. Ε, έχουμε την κρίση η οποία χτυπάει την Ευρώπη και, και με αυτό μπορούμε να πούμε ότι αυξάνονται και διακρίσεις. Α, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λάβει υπόψη της σημαντικού θέματος αυτού που έχει να κάνει με τους Ρώμα. Είχαμε στην αρχή τα πέντε ψηφίσματα που ανέκρινε το Πρακτικό Κοινοβούλιο το 2005. Είχαμε δύο συνόδους κορυφής όπου είδαμε τα θέματα το Ρώμα 2008 και στο Κόρντου το 2010 και συγχαίρω την Ισπανική Προεδρία. Η Επιτροπή επίσης έχει δημοσιεύσει πολλές ανακοινήσεις στο θέμα το Ρώμα και παρακινώντα τι χώρες μέλη να πάρουν πρωτοβουλίε και να υπάρξει μια, ένα συντονισμό, θα λέγαμε, των προσπαθειών τους, ούτω ώστε να ε, περάσουν ουσιαστικά προγράμματα για τους Ρώμα. Ε, από το 2007 έχουν ληφθεί πολλές αποφάσεις και προσπάθειες για να υπάρξει ένταξη των Ρώμα και όλα αυτά ε, δίνουν μια ε, παρότριση, ώστε να συντονιστούν όλες οι ενέργειες. Ε, έχουμε κάποια αποτελέσματα τα οποία μπορούμε να κτυπήσουμε. Υπάρχουν οι κατευθυντήριες γραμμές για να μπορέσουμε να καθορίσουμε τις δράσεις υπέρ των Ρώμα, τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Επίσης, οι κανόνες που έχουν, οι κανόνες που έχουν να κάνουν με το ε, Ταμείο Συνοχής και υπάρχει μια ομάδα εργασία η οποία έχει τεθεί σε εφαρμογή και σε δράση. Επίσης, μια δράση σε μια περίοδο συγκεκριμένη υπέρ των Ρώμα. Έχουμε την Ισπανία και το Βέλιο και την Ουγγαρία που θεωρούν ότι πρέπει να προχωρήσουμε πέρα-πέρα και θα πρέπει να δοθεί μια ένταση, θα λέγαμε, στην κινητικότητα, ούτω ώστε να συντονίσουμε τι πολιτικέ μα. Οι χώρε μέλη έχουν πάρει, αναλάβει κάποιε δεσμεύσει για ουσιαστικά μέτρα για την κοινωνική ένταξη των Ρώμα. Η Βελική Προεδρία κλείνει πλέον και να κάνω ένα μικρό απολογισμό για τις διάφορες δεσμεύσεις και να αναφέρω κάποια σημαντικά θέματα για το μέλλον. Το τρί, η Τρόικα λοιπόν θέλησε οι κοινωνικές δράσεις να δώσουν μια έμφαση στο θέμα το Ρώμα, μια πολιτική mainstream θα λέγαμε και έχει γίνει αυτό σε τρεις διαφορετικές δράσεις. Υπήρξε διάσκεψη για την ε, παιδική ε, φτώχεια το, 2000, το Σεπτέμβριο 2010 και κυρίως για το θέμα δηλαδή των παιδιών το Ρώμα. Πρόσφατα 16-15 Νοεμβρίου που έγινε μια σύνοδο κορυφή στην ε, και το θέμα των διακρίσεων στον χώρο εργασίας όπου δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα που, των ευθυνών που έχουν ε, οι εταίροι, ούτω ώστε να υπάρχει μια συγκεκριμένη ειδική προσέγγιση για του Ρώμα όσον αφορά αυτό το θέμα. Επίση, η διάσκεψη η ευρωπαϊκή για, το, για την συνένεση για τα άτομα που δεν έχουν στέγαση. Και εκεί επίση θίξαμε το θέμα. Υπάρχει μια πτυχή που αφορά με τον προβλεσμό όσον αφορά του Ρώμα. Επίση, η Τρόικα προσπάθησε να διαμορφώσει μια, ένα οδικό χάρτη τους ώστε να γίνουν κάποιες βραχυπρόθεσμες δράσεις. Έχουμε προτάσεις για μια εθνική στρατηγική όσον αφορά την ένταξη των Ρώμα και χαιρόμαστε που θα υπάρχει ένας προγραμματισμός για τον Απρίλιο του 2011. Επίσης θα γίνουν άλλες συνεδριάσεις. Στις Βρυξέλλες έχει προβληθεί κάτι. Αυτό στα πλαίσια πάλι ε, της Προεδρίας της δικής μας, 13 Δεκεμβρίου. Επίσης, μια άλλη δέσμευση τη τροϊκα. Τα, τα διορθωτικά ταμεία να είναι προσβάσιμα στους Ρώμα όσοι έχουν ανάγκη και οι χώρες μέλη να κάνουν σωστά την χρήση αυτών. Επίσης, η Επιτροπή έχει ορίσει μια task force που λέμε, ομάδα κρούση, που αναλαμβάνει να κάνει κάποιες επαληθεύσει αν όντω σωστά γίνεται μια ε, διαχείριση ε, σε σχέση με αυτό το θέμα. Επίσης, να πω, τέλη του 2011 θα έχουμε μια έκθεση και τα συμπεράσματα θα είναι σημαντικά σε σχέση με τις προτάσεις της Ευρώπης για μια ε, συνολική προσέγγιση του θέματος. Επίσης έχουν γίνει πολλές ε, πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εδώ υπάρχει μια προστιθέμενη θα λέγαμε αξία. Και φυσικά τι τίθεται το θέμα της ευθύνης των κρατών μελών. Χρειάζονται φυσικά και πόροι για να γίνει αυτή η δράση. Υπάρχουν ε, αρχές και αξίες οι οποίες στηρίζονται στη χάρτα των θεμελιών δικαιωμάτων και στα πλαίσια της στρατηγικής της Λισαβόνα. Παρ' όλα αυτά η Ρώμα βλέπουμε ότι είναι δαχτυλοδειχτούμενη, είναι απομονωμένη. Επίσης έχουμε την οδηγία η οποία γορεύει τις διακρίσεις σε σχέση με την καταγωγή κάποιου και θα πρέπει να εφαρμοστεί και σίγουρα να προστατευτούν οι Ρώμα. Επίσης το 2009 στη Στοχόλμη είχαμε δει το θέμα που αφορά ε, τις που πρέπει να γίνονται ούτω ώστε να γίνει ένας αγώνας κατά των διακρίσεων και τη ξενοφοβία. Υπάρχει δηλαδή μια τόσο μεγάλη ε, μια έκταση δράσεων όπου δίνεται έμφαση σε αυτό το θέμα διότι οι χώρες μέλη έχουν ένα θα λέγαμε οπλοστάσιο για να μπορέσουν να πολεμήσουν αυτή την πληγή. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει σαφέ ότι δεν θα πρέπει να περιμένει συνεχώ κανεί πρωτοβουλίε νομοθετικέ ή άλλε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσει να προχωρήσει. Χρειάζεται μια θέληση, μια προσπάθεια σε εθνικό επίπεδο και φυσικά να δίνει κανεί και την ετοιμότητα που πρέπει. Στο μέλλον, θεωρώ και με βάση διάφορε συστάσει, χώρε μέλη θα μπορέσουν να έχουν διατάξει οι οποίε θα επιτρέψουν ένα καλύτερο διάρθρωση στο διάλογό του για τα θέματα που αφορούν του Ρώμα σε κάθε χώρα για να μπορέσει κανείς να έχει εθνικές στρατηγικές και δράσεις. Δράσεις δηλαδή που θα είναι καλύτερα προσβάσιμες ή μάλλον προσαρμοσμένες σε κάθε χώρα. Σε βελικό επίπεδο σε σχέση με το διάλογο που κάνουμε με του εκπροσώπους του Ρώμα προτείνουμε ε, όταν θα έχουμε κυβέρνηση, όταν να δούμε πώς μπορούμε να οργανώσουμε κάτι στο Βέλιο ένα όργανο το οποίο να, είναι, να εκπροσωπεί, να είναι επίσημο να εκπροσωπεί τους Ρώμα ε, αυτή την ιδέα θα την υποστηρίξω εγώ. Να έχουμε δηλαδή και επίσης και μια task force σε εθνικό ε, επίπεδο, να γίνουν δράσεις. Κάθε χώρα μέλο δηλαδή θα μπορούσε να έχει μια τέτοια task force για να κάνει τις ανάλογε δράσεις. Είμαστε πεπισμένοι ότι μια πολιτική ένταξη των Ρώμα ε, για να πετύχει πρέπει, πρέπει να γίνει σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά να για να γίνει αυτό θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ε, ανάγκες που έχουν αυτοί οι άνθρωποι, να γίνει σωστή ενημέρωση και να γίνει κατανοητό ότι οι ίδιοι θα πρέπει να συμμετέχουν και στην αξιολόγηση των διαφόρων δράσεων και να μπορέσουν να κάνουν και συστάσεις. Πέρα λοιπόν από όλα αυτά, θεωρώ ότι όσα έχουν να κάνουν με την ε, ανταλλαγή σωστών ε, βέλτιστων πρακτικών ανάμεσα στις χώρες μέλη, είναι σημαντικά όλα αυτά τα θέματα και θα πρέπει να αξιολογηθούν και σωστά. Είναι σαφές λοιπόν ότι υπάρχει μια δέσμευση σε βελικό επίπεδο και δεν σταματάει το ενδιαφέρον του Βελγίου με το τέλος της προεδρίας αυτής. Αλλά θα πρέπει να δούμε στο μέλλον μια προσέγγιση πολύπλευρη με μεγαλύτερη συμμετοχή. Αυτά λοιπόν σαν έναν τρόπο την απολογισμό στα πλαίσια της Βιλικής Προεδρίας. Θα ευχαριστήσω την Επιτροπή Δημόσιων Ελευθεριών που πήραν ε, αυτήν την πρωτοβουλία. Επίσης να πω, ε, συγχαίρω την Ουγγρική Προεδρία που λέει ότι, που έχει αποφασίσει να είναι μία από τις προτεραιότητες Πολύ σημαντική δέσμευση. Επίσης να πω ότι είναι σημαντικό αυτός ο προβληματισμός να μην γίνεται μόνο με λόγο του ότι έχει προκύψει κάτι σε μια χώρα μέλος, αλλά να αποτελεί όντως μια ευρωπαϊκή προτεραιότητα, πολλά μπορούν να γίνουν, πρέπει να γίνουν, ούτω ώστε να αποφύγουμε την περιθωριοποίηση. Όταν βλέπει κανεί την ιστορία, ζουν, βλέπουμε ότι εδώ και δέκα αιώνε ζουν οι Ρώμα στην Ευρώπη. Με τη γλώσσα του, τη λογοτεχνία του, με τη δράση του έχουν συμβάλει στην ευρωπαϊκή ταυτότητα περιθωριοποιώντα λοιπόν αυτού του ανθρώπου, θα λέγαμε ότι περιθωριοποιούμε ένα μέρο τη δική μα ιστορία, του δικού μα πολιτισμού. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ. Εκπροσωπώντα τώρα την επερχόμενη ε, Ουγγρική Προεδρία, ο κ. Ζόλταν Μπαλόγ, υφυπουργό για θέματα κοινωνικών, κοινωνικής ε, ενσωμάτωσης. θα λάβω και εγώ το λόγο στα Ουγγρικά, με επιτρέπετε κυρία Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, αν είμαι εδώ σήμερα μεταξύ σας είναι για να σας μιλήσω εξ ονόματος της νέας Ουγγρικής κυβέρνησης και να σας αναφέρω ποια είναι η θέλησή μας. Η θέλησή μας είναι να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κοινότητα των τσιγκάνων. Αναφέρομαι στους τσιγκάνους και όχι στους Ρώμα, γιατί για μας δεν είναι διάκριση να τους αναφέρουμε ως τσιγκάνους. Ο αγώνας των ε, τσιγκάνων στην Ευρώπη είναι από τα θέματα που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την Ουγγρική Προεδρία. Και εγώ χαίρομαι για το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχει αυτή η προτεραιότητα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το έργο. Γιατί, πρώτα απ' όλα, γιατί πολλοί έχουν αγωνιστεί για να μπορέσει να προχωρήσει αυτός ο αγώνας και να στεφθεί υπό επιτυχία. Η κυρία Λίβια Γιάρογα αγωνίστε εδώ και 10 χρόνια ώστε ο αγώνας αυτός των τσιγκάνων, το Ρωμά, να γίνει κατανοητό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πολλές προσπάθειες λοιπόν για αυτόν τον στόχο και από ανθρώπους που είναι Ρωμά οι ίδιοι και από ανθρώπους που δεν είναι Ρωμά. Υπάρχει επίσης και ένας αγώνας αρνητικού χαρακτήρα γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να αγωνιστούμε για την ενσωμάτιση των Ρώμ, το Ρωμά, αυτό γιατί με τρόπο απαράδεκτο ακόμα και σήμερα εξακολουθούν να υπάρχουν διακρίσεις σε βάρος των τσιγκάνων. Δεν είναι επειδή είμαστε η Ουγγρική Προεδρία που το θέμα το Ρωμά είναι ένα θέμα προτεραιότητος. Ήδη το Μάιο η Ουγγαρία είχε μια νέα κυβέρνηση και αυτή η νέα κυβέρνηση δημιούργησε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και ένα υφυπουργείο που αφορά την ε, ενσωμάτωση των μειονοτήτων και των Ρωμά στην ε, κοινωνία και ιδίω για τα άτομα τα οποία ζουν σε βαθιά ένδια. Μέσα στην Ουγγρική κυβέρνηση λοιπόν έχουμε ένα διαυπουργικό φορέα ο οποίος εργάζεται για να συντονίσει όλες τις ενέργειες που αφορούν τους ε, Ρωμά και που έχει το δικαίωμα αρνησικηρίας σε σχέση με οποιαδήποτε νομοθετική πρωτοβουλία η οποία έχει να αντιμετωπίσει την ένδια των τσιγκάνων, των Ρωμά που ζουν στην Ουγγαρία. Αυτός ο διαυπουργικός φορέας εργάζεται επίσης και, και υπέρ μιας καλύτερης μορφή συντονισμού των πολιτικών της ε, Ουγγαρίας σε σχέση με την κοινωνική ένταξη των μειονοτήτων και το Ρώμα. Έχουμε λοιπόν μια ειδική ανάγκη η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί και υπό το πρίσμα του πολιτισμού, της ε, παιδείας, της υγείας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και φυσικά και της δικαιοσύνης. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αφιερωθούν πόροι και οι πόροι οποίοι είναι διαθέσιμοι θα πρέπει να είναι προσβάσιμοι και προσπελάσιμοι στις κατηγορίες αυτές του πληθυσμού που χρειάζονται αυτή την αρρωγή. Πρέπει να εργαστούμε περισσότερο και να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουμε έτσι να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα στη διάθεσή μας. Είναι πολύ σημαντικό για μας το ότι υπάρχει η δύναμη κρούσης, η ομάδα εργασία αυτή για τους ε, Ρώμα και αναμένουμε να δούμε ποιες είναι οι προτάσεις και οι απαντήσεις που θα δώσει στα προβλήματα αυτά η ομάδα κρούσης αυτή. Όταν έχουμε την πρώτη έκθεση από αυτή την ομάδα στα τέλη του 2010, το Δεκέμβριο 2010, η Ουγγρική Προεδρία θα προβεί στην διατύπωση ενός μη γραφού ενός non-paper που έχει να κάνει με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους Ρωμά στην Ευρώπη. Θα ήταν ενδιαφέρον να υπάρξει λοιπόν και μια μεγαλύτερη δέσμευση των κρατών μέρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βοηθήσουν την κοινωνική ενσωμάτωση των Ρωμά. Γιατί πολλές φορές υπάρχει μια διπλή γλώσσα που είναι ανάγλυφη στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς ακριβώς θα δεσμευτούμε για να δράσουμε Δρούμε επί εθνοτικής βάσης ή δρούμε στον κοινωνικό τομέα. Στην περίπτωση της ε, πλατφόρμας για τους Ρωμά μπορεί να υπάρξουν μια σειρά αποδεσμεύσεις. Παραγματικά χάρη μέχρι το 2020 η Ουγγαρία έχει σαν στόχο να μειώσει κατά 18% τον αριθμό αυτών που ζουν σε απόλυτη ένδια συγκεκριμένα παιδιά ή άτομα τα οποία είναι ε, άνεργοι κτλ. Στην Ουγγαρία σε ένα πληθυσμό 10, 10 εκατομμυρίων η μισή περίπου από αυτούς που ζουν σε βαθιά ένδια είναι Ρωμά, ενώ μόνο 8% των Ούγγρων είναι τσιγκανικής καταγωγής. Και επίσης συνεδητή γλώσσα μιλάμε αφενός για προγράμματα τα οποία βασίζονται στην εθνοτική προέλευση ή για προγράμματα που έχουν οικονομικό-κοινωνικό χαρακτήρα. Στα κρατημέλη λοιπόν και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξουν δράσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπέρ το Ρωμά και τα κράτη-μέλη. Σας έδωσα προηγουμένως και ένα παράδειγμα για ό,τι αφορά τώρα την δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εξετάσει καλύτερα πώς τα διορθωτικά ταμεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς την κατεύθυνση αυτή. Εδώ και πολύ καιρό λέμε ότι πρέπει να υπάρξει μια παρακολούθηση και μια ανάλυση για την χρήση των διαφορετικών πόρων Μέχρι στιγμής όμως είναι μάλλον η εξαίρεση παρά ο κανόνας. Σπάνια ένα πρόγραμμα έχει μεγάλη επιτυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, σε ό,τι αφορά την ανάλυση όλων αυτών των προγραμμάτων θα πρέπει να έχουμε μια κάπως διαφορετική προσέγγιση. για τις διάφορες υποομάδες του πληθυσμού τώρα, τις διάφορες κοινωνικές υποομάδες. Έχουμε να θέσουμε μία σειρά από ερωτήματα. Είναι πραγματικότητα ότι τα κονδύλια τα οποία δίδονται για την ενσωμάτωση φτάνουν πραγματικά μέχρι τις ομάδες στόχους για τις οποίες προορίζονται. Έχουμε εδώ μία ανάλυση του ελεκτικού συνεδρίου της Ουγγαρίας, μία έκθεση η οποία λέει ότι στην πραγματικότητα πολύ λίγα από τα κονδύλια τα οποία έχουν αφιερωθεί στους Ρωμά έχουν πράγματι φτάσει τους τελικούς αποδέκτες. Δεν έχουμε εξάλλου και επακριβή στοιχεία στατιστικά σε σχέση με το βαθμό χρησιμοποίησης από τους Ρωμά των κονδυλίων αυτών που αφορούν αυτούς τους ιδίους. Πρέπει επομένως να εργαστούμε περισσότερο για να δημιουργήσουμε και ένα σύστημα αξιόπιστων <clears throat> δικτών στην Ευρώπη που θα μας επιτρέψουμε, επιτρέψουν να καταλάβουμε καλύτερα πώς χρησιμοποιήθηκαν τα ποσά υπέρ των Ρωμά και μια σειρά από δείκτες που θα μας δώσουν καλύτερες κατευθύνσεις για να ευνοήσουμε την, την μεγαλύτερη χρησιμοποίηση αυτών των κονδυλίων από τους ε, Ρωμά. Και εξάλλου θα πρέπει να υποχρεωθούν τα κράτη-μέλη να συντάσσουν εκθέσεις οι οποίες θα έχουν να κάνουν με την εφαρμογή των μέτρων τα οποία έχουν αποφασιστεί υπέρ των Ρώμα. Μέσα στα πλαίσια του Συμβουλίου εμείς θα αντιμετωπίσουμε μία σειρά από νομοθετικές προτάσεις και όπως ελέγχθη στις 8 Απριλίου του 2011 θα λάβει χώρα στη Βουδαπέστη και η πλατφόρμα για τους Ρωμά. και όπου θα αντιμετωπιστούν επίσης και περαιτέρω ερωτήματα σε σχέση με το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρωμά. Έχουμε λοιπόν αυτό το ραντεβού για τις 8 Απριλίου στη Βουδαπέστη. Και τον Απρίλιο και τον ε, Ιούνιο θα έχουμε συνεδριάς του, του Συμβουλίου Υπουργών για την Παιδεία και συμβούλιο, το συμβούλια Υπουργών ε, Απασχόλησης και το Συμβούλιο Εσωτερικών και Δικαστικών Θεμάτων θα αντιμετωπίσει και αυτό τα ζητήματα αυτά. Με την συνεργασία αυτών των Συμβουλίων πιστεύουμε λοιπόν ότι θα μπορέσει να αρθρωθεί καλύτερα αυτή η στρατηγική και αν όλα πάνε καλά μπορούν να υπάρξουν συγκεκριμένε και απτές συστάσεις προς τα κράτη-μέλη. Μια ακόμα φορά υπάρχουν και κάποιες εσωτερικές αντιφάσεις σε όλη αυτή τη διαδικασία. Πιστεύουμε ότι η ενσωμάτωση των Ρωμά θα πρέπει να γίνει με το έργο των κρατών μελών. Συγχρονώς όμως υπάρχει μια ευρωπαϊκή διάσταση αυτής της κοινωνικής ένταξης των Ρωμά. Υπάρχει αυτή η ευρωπαϊκή διάσταση γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να αντιμετωπίσουμε θέματα όπως η οργανωμένη εγκληματικότητα. Θα πρέπει να εργαστούμε από κοινού για να δώσουμε τη δυνατότητα να εξασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία όλων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεν, αλλά χωρίς αυτό το δικαίωμα να την χάνει χειραγώγησης και εκμετάλλευσης από εγκληματίες, από εγκληματικά στοιχεία. Πρέπει να υπάρχουν και κάποια λοιπόν εμπόδια για την ελεύθερη κυκλοφορία. Γιατί πολλές φορές τα θύματα αυτής της μεγάλης εγκληματικότητας είναι και αυτά ανήκοντα στην κοινότητα των Ρωμά. Είμαι σίγουρος λοιπόν ότι αυτό ισχύει και για την Ουγγαρία και για άλλες χώρες της Ευρώπης, ότι ανεξάρτητα από τη φύση των προβλημάτων θα πρέπει να βρούμε τους τρόπους να λύσουμε τα προβλήματα αυτά. Ο τρόπος για μένα αυτός είναι να πείσουμε την πλειοψηφία των πολιτών μας ότι η προσέγγιση μας είναι η σωστή. Γιατί πολλές φορές η πλειοψηφία των πολιτών αγνοεί το θέμα της ενσωμάτωσης στο Ρωμά. Δεν πρέπει να λησμονήσουμε ότι πολλοί στην Ευρώπη έχουν προκαταλήψεις εναντίον του Ρωμά. Ποιο λοιπόν θα είναι το κλειδί της επιτυχίας στον τομέα αυτό. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί αυτή η ενσωμάτωση στο Ρωμά, όχι μονάχα για λόγους ηθικής και αλληλεγγύης, αλλά και γιατί είναι προς το συμφέρον όλων να έχουν ενσωματωθεί οι Ρωμά στην κοινωνία και να απολαμβάνουν και αυτοί των ίδιων δικαιωμάτων που έχουν και όλοι οι άλλοι πολίτες στις κοινωνίες μας. Από οικονομική έποψη έχει καταδειχθεί ότι ο αποκλεισμό σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο είναι πολύ πιο πολυδάπανος από την αποτελεσματική ενσωμάτωση και την ε, εξάλληψη των διακρίσεων. Η Ουγγαρία έχει γνωρίσει το θέμα των Ρωμά σε σημαντική έκταση. Πολλές φορές αντιμετωπίζει κανείς στην Ουγγαρία με ποδοσφαιρικό τρόπο, δηλαδή όλοι ξέρουν τι είναι το ποδόσφαιρο, όλοι μιλάνε για το ποδόσφαιρο χωρίς να ξέρουν πολλά πράγματα. Στην Ουγγαρία λένε πολλοί ότι έχουμε τσιγκάνους στη χώρα μας, αλλά κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς είναι αυτοί οι άνθρωποι και ποια είναι τα προβλήματα τα οποία τους απασχολούν. Και εγώ μπορώ να επαναλάβω αυτά τα οποία είπε η κυρία Μιλκέ, ότι πρέπει καταρχήν να υπερασπιστούμε τις αξίες μας, τις εθνικές και τις ευρωπαϊκές στον τομέα του Ρωμά. Σας ευχαριστώ κύριε Μπαλόγ. Ερχόμαστε τώρα στη φάση ερωτήσεων και απαντήσεων με κάποια καθυστέρηση. Έχω πολλούς συναδέλφους οι οποίοι ζήτησαν το λόγο και επίσης και συμμετέχοντες στο, στα πάνελ που θέλαν να λάβουν το λόγο. Θα είμαι ιδιαίτερα αυστηρή, θα ζητήσω καταρχήν από τα μέλη των Επιτροπών να είναι ιδιαίτερα σύντομοι. Μήπως μπορείτε να σιωπήσετε, μήπως μπορείτε να κάνετε ησυχία, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε αλλιώς. Πρώτα θα δώσω το λόγο στα μέλη και σας παρακαλώ να είστε ιδιαίτερα σύντομοι, το πολύ ένα λεπτό, ένα ενάμιση λεπτό. Και στη συνέχεια θα καλέσω όλους τους ε, άλλους συμμετέχοντες οι οποίοι θέλουν να λάβουν το λόγο. Δεν δέχομαι λοιπόν άλλες αιτήσεις. Έχω κλείσει τον κατάλογο των ερωτώντων. Η κυρία Βέμπα έχει το λόγο καταρχήν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Λίβια που οργάνωσε την ακρόαση αυτή. Θα προτιμούσα να ήμασταν στην πρωινή αίθουσα συνεδρίασης που ήταν μεγαλύτερη. Θα χωρούσαμε καλύτερα. Όσον αφορά αυτά που συζητήθηκαν, νομίζω ότι βρισκόμαστε σε σημείο όπου εμείς ως βουλευτές, ευρωβουλευτές, θέλουμε να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα. Δεν είναι ώρα για ανταγωνισμό μεταξύ μας. Δεν είναι ώρα να δείξουμε ποιος είναι πιο έξυπνος από τον άλλον, είναι ώρα να συνεργαστούμε εάν θέλουμε να πετύχουμε ε, συγκεκριμένα αποτελέσματα. Υπό το φως αυτό πιστεύω ότι ό,τι τροπολογίες υποβληθούν για την έκθεση της Λίβια θα πρέπει να είναι στο πνεύμα ε, μιας επικοδομητικής πρόσβασης και που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από την Κομισιόν όταν αυτή εκπονήσει το δικό της έγγραφο. Δεν τολμώ να στρατηγική. Ταυτόχρονα θα πρέπει να πω ότι χαίρομαι πολύ με πολλά από τα πράγματα που κάνει εδώ και καιρό η κυρία Ρέντιν και που ανέφερε σήμερα. Επιμένει στην ελεύθερη κινητικότητα και πιστεύω ότι ως μέλος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η ελεύθερη κινητικότητα και κυρίως ε, η παραβίασή της. Αρκεί να ανάψει κανείς την τηλεόραση να δει τι γίνεται αυτές τις μέρες στη Λιόν. Που πετάνε τον κόσμο στο δρόμο. Άσχετα από το ότι χιονίζει, είναι χειμώνας ε, κτλ. Ε, αυτό δεν ενδιαφέρει καθόλου τις γαλλικές αρχές. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να στηρίξουμε την Επίτροπο Ρέντινγκ στο θέμα αυτό. Ταυτόχρονα σήμερα μας παρουσιάστηκε μια νέα έννοια, το νέο ε, πλαίσιο για τις εθνικές στρατηγικές ε, για την ένταξη των Ρώμα. Ε, αυτό είναι νέο, χρειάζομαι χρόνο να το χωνέψω, αλλά νομίζω ότι θα είναι σημαντικό να έχουμε μια νέα συνάντηση με την Επίτροπο. Θα χρειαστούμε διευκρινήσεις για το θέμα αυτό και θα πρέπει αυτό να γίνει πριν τον Απρίλιο του 2011. Θα πρέπει να καταλάβουμε καταρχήν, θα πρόκειται να υπάρξει η ανακοίνωση από την Κομισιόν, ε, το Κοινοβούλιο θα υποβάλει το δικό του ψήφισμα, ποιες ε, θα είναι οι οικονομικές συνέπειες για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, για τον προϋπολογισμό των κρατών μελών, ποιος θα είναι ο νομικός χαρακτήρας της πρότασης αυτής απέναντι στα κράτη-μέλη. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζουμε τι θα γίνεται με τι θα γίνει με τα benchmarks και τη χρηματοδότηση. Εάν μπορεί ε, κάποιο από την Κομισιόν να αποπαντήσει, θα χαρώ πολύ, αλλά εγώ θα πρότεινα ε, μια ε, νέα συνάντηση. Ε, η πρόεδρο διακόπτει την ομιλήτρια. Ναι, συγχωρήστε με, αλλά τώρα που μιλάμε για του Ρώμα και του Τσιγκάνου, πρέπει να υποβάλω ένα τέτοιο αίτημα, διότι θέλω να πιστεύω ότι η Ουγγρική Προεδρία θα καταλάβει ότι Το θέμα των Ρώμα απαιτεί πολιτική βούληση να δείξουμε κάτι. Αν τα κράτη-μέρη το δεχτούν αυτό, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση το δεχτεί αυτό και το ε, δικαστήριο και το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πιστεύω ότι ε, θα πρέπει και η Προεδρία να συνεχίσει να ασχολείται με το θέμα των Ρώμα. Ευχαριστώ one minute or one and a half minute. Otherwise we... Ένα, ενάμιση λεπτό, αλλιώς, ένα, ενάμιση λεπτό το πολύ, αλλιώς δεν θα προλάβουμε. Ο κύριος Σούγκορ έχει το λόγο. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος γιατί ο υπουργός, ο κύριος Μπάλοκ ανέφερε ήδη αυτά που ήθελα να πω εγώ. Πρέπει να εξασφαλίσουμε την ενσωμάτωση σε επίπεδο ευρωπαϊκών αρχών. Πολλές φορές ε, υπάρχουν προβλήματα αντιμετώπισης μειονοτήτων και μη αποδοχής διαφορετικών κοινωνικών και εθνοτικών ομάδων που καταδεικνύουν ότι κάποια κράτη-μέλη θα πρέπει πραγματικά να αποδεχτούν τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες που δεν το έχουν πράξει πλήρως. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, voi fi foarte scurt. Πολύ σύντομα. Ε, καταρχήν, αφότου άκουσα όλους τους προλαλήσαντες, ξαφνικά ε, αποκτώ ένα, μια αισιοδοξία για το μέλλον. Επιτέλους ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι σωστό για αυτήν την κοινότητα. Αυτό που θα μπορούσα να πω είναι η κυρία Γιαννιούκα, η συγγήτρια, έχει συντάξει ένα σχέδιο έκθεση καταπληκτικό. Και φυσικά θα υπάρξουν και τροπολογίες. Φυσικά καταλαβαίνει κανεί ότι δεν κάνουμε ένα ολόκληρο μισθόριμα. Γιατί όμω, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Παρ' όλα αυτά έχω μια αισιοδοξία, διότι ακούσαμε και την Επίτροπο κυρία Ρέντινγκ, η οποία επιμένει ότι η ένταξη, η ενσωμάτιση των Ρώμα θα πρέπει να είναι θέμα ευρωπαϊκού επίπεδου για όλη την Ευρώπη και να δεσμευτούν όλε οι χώρε μέλη. Και τέλο, ε, θα ήθελα να πω ότι Διαπιστώνω επίσης μετά από αυτά που άκουσα ότι τα προβλήματα που έχουν η Ρουμανία, η Ουγγαρία και άλλες χώρες όπου υπάρχουν κοινότητες στον Ρώμα είναι ανάλογα προβλήματα. Υπάρχουν μικρές διαφορές έλεγα. Η ουσία είναι πάντα ίδια όλων αυτών των προβλημάτων. Ευχαριστώ. Τέσσερα θέματα. Καταρχήν ένα... Σα ευχαριστήσω διότι σιγά σιγά προχωράμε σε πιο συγκεκριμένα θέματα και πιστεύω θα καταλήξουμε σε μια πολύ καλή έκθεση. Θα ήθελα να ε, πω αυτό καταρχήν. Δεύτερον, για μένα είναι πολύ σημαντικό κατά την ανάπτυξη της στρατηγικής αυτής τα κράτη-μέλη να δεσμευτούν να δεσμευτούν ε, ε, με συγκεκριμένες υποχρεώσεις από τις οποίες να μην μπορούν να ξεφύγουν με δικαιολογίες. Είναι Πολύ σημαντικό αυτό, διότι μπορούμε να λάβουμε ό,τι αποφάσεις θέλουμε, εάν δεν ε, καταφέρουμε στα κράτη-μέλη να υλοποιηθούν αυτά, τότε θα αποτύχουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Επίσης, όσον αφορά την ε, χρηματοδότηση και τη χρήση πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι δυνατόν να μην απορροφούνται οι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το αναφέρατε. Θα πρέπει να σκεφτούμε μήπως θα πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε για κυρώσεις. Τη στιγμή που δεν απορροφούνται τέτοιοι πόροι που είναι πολύ σημαντική η χρήση τους για να αποφευθούν οι διακρίσεις. Επίσης, ε, η ζωή των Ρώμα είναι, διαφέρει πολύ από τόπο σε τόπο εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν μιλάμε λοιπόν για τους Ρώμα θα πρέπει να φροντίσουμε να, φροντίζουμε, να έχουμε υπόψη μα ότι στα 12 αυτά εκατομμύρια ανήκουν και άνθρωποι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, που δεν πρέπει να τους ξεχάσουμε τελείως. Και πραγματικά δεν μου αρέσει ο όρο τσιγκάνη. Στη Γερμανία ο όρος αυτός ε, είναι δείγμα διάκρισης. Και θα είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα για μας, αν μιλάμε για τσιγκάνους. Τελευταία πρόταση, πραγματικά τελευταία πρόταση θα πρέπει οι μη κυβερνητικέ οργανώσει και οι κοινότητε στον Ρώμα να συμμετέχουν στην όλη διαδικασία. Αυτό είναι το Α και το Ω. Μπορούμε να λάβουμε ό,τι αποφάσει θέλουμε. Χωρί του Ρώμα δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Του χρειαζόμαστε από την πρώτη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σε δύο λεπτά λυπάμαι, αλλά είναι πολύ δύσκολο να καλύψει κανεί όλη τη θεματολογία. Πρέπει να πω ότι στη χώρα μου η οι τσιγκάνοι χαίρονται, έχουν περηφάνεια που μπορούν να ονομάζουν τον εαυτό τους τσιγκάνο. Και επομένως υπάρχει προκατάληψη εναντίον των ε, ορισμένων ονομασιών. Για μένα αυτό είναι, είναι μια από τις πρώτες συζητήσεις που πρέπει να κάνουμε για το θέμα της ονομασίας. Κύριε Υπουργέ, για την ε, κοινωνική ενσωμάτωση. Επειδή θα επανέλθουμε στην Ουγγρική Προεδρία για το θέμα αυτό και επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, θέλω να σταθώ σε δύο θέματα. Όταν μιλάμε για τον, για τον πληθυσμό των τζιγκάνων και για την κουλτούρα των Ρωμανί και συγχρόνω μιλάμε για εγκληματικότητα στην Ευρώπη, δεν κάνουμε τίποτα, δεν προχωράμε. Εξακολουθούμε να έχουμε την ίδια κατηγοροποίηση. Οι, οι εγκληματίες, οι κακοποίοι έχουν συγκεκριμένη, συγκεκριμένο όνομα και επίθετο. Δεν είναι υποχρεωμένοι να ανήκουν στους τσιγκάνους, μπορούν να ανήκουν και στους μη τσιγκάνους. Δεν μπορούμε επίσης να μιλάμε για τον πληθυσμό Ρωμανί. Όταν μιλάμε έτσι για τους ανθρώπους αυτούς, ήδη τους στιγματίζουμε, ήδη τους χαρακτηρίζουμε με έναν τρόπο. Αυτό λοιπόν είναι μια πρώτη στη πτυχή. Δεν πρέπει να συνδέουμε την εγκληματικότητα με τους Ρωμανί, με τους ε, Ρωμά. Δεν μπορούμε λοιπόν να έχουμε μια τέτοια αντιμετώπιση όταν θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα είναι πλήρη μέλη της κοινωνίας μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και μια δεύτερη ιδέα που θέλω να τονίσω είναι να, ότι είναι αδύνατο να ξέρει ακόμα η Ουγγαρία αν έχουν φτάσει σε αυτούς τα κονδύλια, στους Ρωμά τα κονδύλια τα οποία έχουν δοθεί για αυτούς. Εδώ υπάρχει πραγματικά μια ευθύνη ενός κράτους να ξέρει πού πηγαίνουν τα χρήματα αυτά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δώσει κάποια χρήματα, αλλά αυτά τα χρήματα είναι υποχρεωτικό να φτάσουν στην ομάδα στόχου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι απαραίτητο να εξασφαλίσει ότι θα προχωρήσουν αυτοί οι άνθρωποι προς την κατεύθυνση του να γίνουν πλήρεις πολίτες. Αν δεν έχουν λοιπόν εκμεταλλευτεί αυτά τα ποσά, αυτό είναι πραγματικά κρίμα, γιατί στη δική μου χώρα έχουν δοθεί πάρα, πολύ, πάρα πολλά ποσά προς την κατεύθυνση αυτή και δεν υπάρχουν ούτε προκαταλήψεις ούτε αποκλεισμό κοινωνικό. Είναι όπω όπως όλοι οι άλλοι και έχουν πάρει κονδύλια του κοινωνικού ταμείου όπω οποιοδήποτε άλλο πολίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρία Μπόσκου, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Δύο σημεία θα θίξω. Το δικ... Για τα 12 εκατομμυρίων Ευρωπαίων. Το θέμα έχει να κάνει με την ασφάλεια. Ε, από τότε που είδαμε όλες αυτές τις ε, δράσεις εναντίον των Ρώμα υπάρχει κάποιος φόβος ότι, ότι υπάρχει μια πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο που στρέφεται κατά αυτών και κρίμα που η Επιτροπή δεν ε, έδραξε αυτή την ευκαιρία για να καταπολεμήσει τις διακρίσεις αυτές. Ελπίζω ότι χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι να νιώσουν μια ασφάλεια. Ε, επίσης, έχουμε να κάνουμε το, το δεύτερο θέμα τώρα, το οποίο έχει να κάνει με την ενσωμάτιση αυτών των ανθρώπων. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η άποψη των εισηγητών. Όλοι δεν είναι παρόντες. Αναφέρομαι στην ενσωμάτιση την πολιτιστική αυτών των ανθρώπων, 12 εκατομμύρια άνθρωποι που έχουν δική τους πολιτιστική παράδοση. Συχνά έχω, έχει κανείς την εντύπωση ότι ζητεί από αυτούς να ενσωματωθούν, να φανιστούν να, κατά κάποιο τρόπο, να χάσουν την ιδιαιτερότητά τους. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω ποια είναι η θέση των εισηγητών πάνω σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ehm, Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομο. Θεωρώ υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Όταν μιλάμε δηλαδή για δικαιώματα, αλλά ξεχνάμε το θέμα των υποχρεώσεων. Όλοι σίγουρα συμφωνούμε ότι υπάρχουν μεγάλα προβλήματα. Ότι η κοινότητα των Ρώμα ε, αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα στις διάφορες χώρες μέλη. Ε, προβλήματα μπορούν να αποφευθούν. Αλλά θα πρέπει να είμαστε σαφείς λέγοντας ότι, ότι η συμπεριφορά αυτής της κοινότητας δημιουργεί πολλά προβλήματα. Για παράδειγμα, όταν δημιουργούνται ε, κατασκηνώσεις σε, χώρες, σε χώρους δεν επιτρέπεται, υπάρχει ένα πρόβλημα. Βλέπουμε επίσης ότι ε, πώς παροτρύνονται τα παιδάκια από τους γονείς να, κάνουν, να ζητιανεύουν. Δεν τα λέμε αυτά. Μόνο σκεφτόμαστε τα, για τα αρνητικά στοιχεία, ε, αλλά πρέπει να θίξουμε και την άλλη πλευρά. Τρεις ιδέες. μονάχα. Καταρχήν, τα δικήματα δεν διαπράττουν κοινότητε, τα διαπράττουν άνθρωποι. Αυτού του ανθρώπου θα πρέπει να διώξει κανεί, όχι μια ομάδα ανθρώπων. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, νομίζω ότι είναι σημαντικό και υπογραμμίζω αυτό που είπε η κυρία Ρομέρο, το θέμα τη ονομασία, τη έννοια. Τσιγκάνι, Ρώμα, όλα αυτά. Καλό είναι να έχουμε μια ονομασία η οποία να μην δημιουργήσει προβλήματα στην χρήση της, αλλά και επί τη βάση του ότι έχει αποδοχή σε ορισμένε περιοχές και ορισμένε κοινότητε. Τρίτον, πολλές φορές έχουμε θίξει το θέμα της ελευθερίας κυκλοφορίας. Και πιστεύω ότι εδώ χρειάζεται μια απόλυτη σαφήνεια. Δεν πρόκειται μονάχα για ελεύθερη κυκλοφορία, είναι και ένα θέμα διάκρισης. Και εδώ νομίζω ότι αυτό το οποίο χρειάζεται και από την πλευρά της Κομισιόν είναι να αντιμετωπίσει την έννοια της διάκρισης. Γιατί έχει αντιμετωπίσει το θέμα αποκλειστικά και μόνο από την πλευρά της ελεύθερη κυκλοφορίας και όχι της διάκρισης που για μένα είναι πιο σημαντική. Τέταρτο και, σημαντική, τελευταίο σημείο. Μιλάμε όχι για μια μειονότητα στην Ευρώπη, αλλά για Ευρωπαίους πολίτες και πολίτησες. Αυτό πρέπει να είναι το σημείο το οποίο πρέπει να είναι η κίνησή μας αν θέλουμε με πατερναλιστικό τρόπο να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα μια μειοψηφία, δεν θα καταλήξουμε πουθενά. Αν ξέρουμε ότι μιλάμε για πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, από εδώ και πέρα μπορούμε να έχουμε μια σοβαρή συζήτηση. Thank you. Ευχαριστώ. Πηγαίνω στους πέντε επόμενους ομιλητές, οι οποίοι θέλουν να λάβουν το λόγο και θα είμαι πάρα πολύ αυστηρή και μετά από ένα λεπτό θα σας κλείσω το μικρόφωνο η κυρία Μιράντα Βολασέντο από το Φινλανδικό Φόρουμ των ε, Ρωμά. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο κυρία Πρόεδρε. Ε, θέλω να ευχαριστήσω και την κυρία Λίβια Γιαρόκα για την ε, καλή δουλειά που έχει κάνει και την πρόκληση που, με την οποία έχει αποφασίσει να ασχοληθεί. Καταρχήν, όταν μιλάμε για τους Ρώμα και τη στρατηγική των Ρώμα, άκουσα σήμερα εδώ πολλούς ομιλητές που μιλάνε για ευρωπαϊκή στρατηγική, ευρωπαϊκό πλαίσιο, ε, για, την, για, την, ε, για τους Ρώμα. Όποιο και να είναι το όνομα, χρειάζεται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο κάτι τέτοιο. Και επίσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς θα φροντίσουν να συμμετέχουν οι ίδιοι οι Ρώμα στη διαδικασία αυτή, διότι ό,τι στρατηγική πολιτική και να έχετε, εάν αφήσετε απ' έξω τους ε, Ρώμα και είναι απλά πάλι στόχος διαφόρων πολιτικών χωρίς να ε, καταλαβαίνουν ε, τι γίνεται και να ε, συμμετέχουν εκεί οι ίδιοι ώστε να αφοσιώνονται στον ίδιο στόχο, αυτό είναι είναι πολύ σημαντικό να γίνει. Αυτό να το έχετε κατά νου, ό,τι στρατηγική και αν ε, έχετε στόχο να ε, προγραμματίσετε. Θα είμαι σύντομο. Εγώ μιλάω εδώ με την ιδιότητα τη δημάρχου μια περιοχή που έχει πολλά προβλήματα. Εγώ για πρώτη φορά λαμβάνω μέρο σε μια συνεδρίαση σαν και αυτή και ακούω σημαντικά πράγματα. Παρά όλα αυτά να σας πω ότι αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα και διότι έχουμε προβλήματα τα οποία τα αντιμετωπίζουμε όχι όπως κάνετε εσείς ε, συζητάτε τα θέματα εδώ ε, σε αυτήν την αίθουσα. Ε, εδώ έχουμε να κάνουμε μια εμπειρία στο χώρο στον οποίο γίγονται τα ε, προβλήματα αυτά. Υπάρχουν διαφορές από χώρα σε χώρα. Ε, θα είμαι σύντομη αυτό που θεωρώ εγώ είναι ότι η, η, ο Δήμος θα πρέπει να κάνει μια προσπάθεια να ενσωματώσει τους ε, Ρώμα. Θα πρέπει να κληθούν αυτοί εδώ διότι οι, δήμα, οι Δήμοι στις Μαρχίες είναι αυτοί που ξέρουν καλύτερα αυτά τα προβλήματα. Συγγνώμη έτσι μιλάω γρήγορα γρήγορα γιατί μου δώσατε μόνο ένα λεπτό. Υπάρχουν λοιπόν όλα αυτά τα προβλήματα, ε, υπάρχουν σχέδια μέσω και βράχη πρόθεσμα και να σας πω Φέρει πει, μια οικογένεια που έχει 5, 10, 15 παιδιά. Τε, οι γονεί δεν ασχολούνται με το αν θα πάνε τα παιδιά στο σχολείο. Δεν έχουν δουλειά, πει. Και η, κυβέρνηση να ασχολείται ε, με το θέμα τους. Στη Ρουμανία, παράδειγμα, είναι εγκαταλειμμένοι οι Ρώμα. Πώς θα ενδοματωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Μπορεί λοιπόν κανεί να κάνει κάποια σχέδια. Οι γονεί δεν έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν. Μια στιγμή, μια στιγμή, ακόμα, κύριε Πρόεδρε. Έδωσα ένα παράδειγμα απλώ. Και να σας πω την άποψή μου. Θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουμε ε, σχέδια τα οποία να είναι βραχυπρόθεσμα για πολυμελείς οικογένειε. Θεωρώ ότι τα κονδύλια που έχουν διατεθεί μέχρι τώρα δεν είναι κονδύλια τα οποία έχουν φτάσει στο στόχο τους. Για, δηλαδή ουσιαστικά προβλήματα. Ορισμένα κονδύλια ε, δεν καταλήγουν εκεί στο στόχο τους και τα απαραίτητα σχέδια που μπορούν να αντιμετωπίσουν προβλήματα δεν ολοκληρώνονται. Council Well, thank Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο, κυρία Πρόεδρε. Και σας ευχαριστώ για την διοργάνωση αυτής της ε, συζήτησης και για την πρόσκληση προς το Συμβουλίο της Ευρώπης. Έχουν ζητήσει πολλοί να ληφθούν υπόψη τα συγκεκριμένα μέτρα. Και εγώ μπορώ να σας δώσω ήδη μια τέτοια πρόταση που είναι και μία από, τη, από τα πορίσματα της συνάντησης υψηλού επίπεδου που έγινε στο Στρασβούργο στις 10 Οκτωβρίου μετά από τα γεγονότα που έλαβαν χώρα σε διαφορές χώρες της Ευρώπης τα εφέτος. Οι εκπρόσωποι και των 47 μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης που περιλαμβάνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκπρόσωποι της κοινότητας των Ρωμά συναντήθηκαν. Ένα από τα συμπεράσματα, κυρία Πρόεδρε, είναι ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τους λεγόμενους μεσολαβητές Ρωμά, που θα δώσουν νομική και διοικητική αρρωγή και συμβουλές στις κοινότητες των ε, Ρώμα. Μπορεί να είναι Ρωμά, μπορεί να είναι ε, αστυνομικοί, εκπαιδευτικοί, άτομα που είναι κοινωνική βοηθή και τα λειτουργεί κτλ. Θα εκπαιδευτούν από το Συμβούλιο της Ευρώπης 440 τέτοιοι μεσολαβητής, αλλά μπορούμε να φτάσουμε μέχρι 1.400. Και εδώ τίθεται ένα θέμα χρηματοδότησης και πόρων. Επομένως, εναπόκειται σε εσά αν θέλετε να εμπλακείτε. Και επίσης υπάρχει ένα αντίστοιχο πρόγραμμα εκπαίδευσης για δικηγόρους οι οποίοι ειδικεύονται σε περιπτώσεις που εμπλέκονται Ρωμά. Το αφήνω στην κρίση σας. Ευχαριστούμε κύριε Πρέσβη. Ο κύριος Μπόρς, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Κύριε Μπάσου, έχετε το λόγο. Δεν ζήτησα το λόγο, ξέρετε. Μου τον δίνετε. Τι να πω. Αν θα χρειαζόταν να πω κάτι σε σχέση με αυτά που ακούστηκαν, ε, θα μιλήσω και αύριο. Εμείς χρειαζόμαστε μια ε, διαδικασία, μια διαφάνεια στο πώς χρησιμοποιούνται τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει αυτό όχι μόνο αρχές ευρωπαϊκές αλλά υπάρχουν και μη κυβερνητικέ οργανώσεις και οι χρήστες να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία διότι θα βρισκόμαστε πάντα στην ίδια κατάσταση. Δηλαδή, κανεί, όπω και σήμερα, δεν θα ξέρει τι ακριβώ γίνεται με τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Παράδειγμα στη Βουλγαρία. Φτάνουν κονδύλια, αλλά κανεί δεν ξέρει πού βρίσκονται αυτά τα κονδύλια, πού καταλήγουν. This uh, from the Ευχαριστώ κυρία Φαντάτσι. Θέλω ευχαριστήσω καταρχήν την κυρία Γιαροκά για την ευκαιρία που μας έδωσε να είμαστε όλοι εδώ. Εγώ εκπροσωπώ το, την ε, ομάδα Ρομ Ευρώπη πάνω από 40 φορείς εθνικού και τοπικού χαρακτήρα. Έχουμε καμιά εικοσαριά επιτροπές στήριξης οι οποίες δρούν σε καθημερινό επίπεδο για να βοηθήσουν τους μετανάστες, τους Ρωμά στην Γαλλία. Αγωνιζόμαστε για το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων αυτού του πληθυσμού και την εξασφάλιση των δικαιωμάτων τους και έχουμε μία αρκετά ανησυχητική διαπίστωση στην κατάσταση στη Γαρία μετά από τα γεγονότα του καλοκαιριού δεν άλλαξε απολύτως τίποτα. Ακούσαμε την Επίτροπο, την κυρία Ρέντιν, η οποία είπε ότι η Γαλλία έδωσε εγγυήσεις για τη δυνατότητα να σεβαστεί το κοινοτικό δίκαιο. Σήμερα βλέπουμε τις προτάσεις για τροποποίηση του νόμου για την ε, μετανάστευση και την ασφάλεια που στρέφονται κατά του κοινοτικού δικαίου. Δεν υπάρχει καμία διαφάνεια σε σχέση με αυτέ τι υποθέμενες εγγύησει που δόθηκαν στην κυρία Ρέν. Επίση, η πολιτική της Γαλλίας βασίζεται στον αποκλεισμό των ε, Ρωμά και στην ε, πρόθεσή τους προς τις χώρες προέλευσής τους. Εμείς αναρωτιόμαστε πώς επί τη βάση αυτή μπορεί η Γαλλία να αναπτύξει προγράμματα συμπερίληψης και ένταξης των Ρωμά. Ευχαριστώ πολύ. Θα ζητήσω από τον κύριο Μπαλό να απαντήσει στα ερωτήματα αυτά και να αντιδράσει και μετά θα ζητήσω από την εισηγήτρια να επανέλθει στα θέματα τα οποία τέθησε. Κύριε Μπάλοκα, έχετε το λόγο. Αν μου επιτρέπετε, θα Ίσως ε, θα, θα είμαι πιο σαφής γιατί πολλά εξαρτώνται από την ε, γλώσσα και την κατανόηση της γλώσσας. Είναι πολύ σημαντική η χρήση της γλώσσας όταν μιλάμε για τέτοια προβλήματα. Μπορεί κανείς να προσπαθήσει να μιλήσει με μια αποστηρωμένη γλώσσα, η οποία δεν οδηγεί σε παρεξηγήσεις, αλλά δεν οδηγεί και σε μια κατανόηση για την κατάσταση των ανθρώπων με τους οποίους απασχολούμαστε σήμερα. Δεν νομίζω ότι είναι χρήσιμο να μιλάμε για ονομασίες και προσδιορισμούς θεωρώ ότι αυτή η άποψη για τους ε, τσιγκάνους που έτσι κι αλλιώς δεν είναι ακριβώς η διαχρήση της ε, λέξης τσιγκόινερ στη Γερμανία ότι είναι ίσως λιγάκι ατυχή, ατυχής. Αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δίνουν το όνομα αυτό στους εαυτούς τους, αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ο αυτοπροσδιορισμός ότι είναι βάση μιας ε, διάκρισης. Όταν υπάρχει λοιπόν ένα σύστημα αυτοδιοίκηση των Ρωμά που του ονομάζει τσιγάνους παραδείγματο χάρη, αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το αποδεχτούμε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν ένα αλλάξ τι έννοια τσιγάνος και Ρωμά. Αυτό είναι αποδεκτό στην ε, Ρουμανία. Το βασικό είναι να αναφέρεται ο προσδιορισμός αυτός με σεβασμό και όχι με περιφρόνηση. Νομίζω ότι μπορούν να τύχουν αξιοπρεπούς αντιμετώπισης και οι τσιγάνοι και οι Ρωμά επί τη βάση μιας ονομασίας. Τώρα για τη στρατηγική πλαίσιο, για την εθνική στρατηγική, για τη στρατηγική των Ρωμά, για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δική μου κατανόηση είναι ότι η Κομισιόν θα προετοιμάσει μία ανακοίνωση η οποία θα αποτελέσει και το πλαίσιο για τις ε, <clears throat> επιμέρους εθνικές στρατηγικές για τη συμπερίληψη των Ρωμά οι οποίε θα αποκτήσουν σάρκα και οστά στα κράτη-μέλη και με τι προσπάθειες των κρατών μελών. Αυτές αυτή η ανακοίνωση λοιπόν της Κομισιόν, αυτό το κείμενο πλαίσιο, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και από τα επιμέρους ε, ε, συμβούλια υπουργών, τα οποία θα πρέπει να συζητήσουν το θέμα αυτό. Για τα θέματα της χρηματοδότηση, Για την οργή ορισμένο ότι τα χρήματα αυτά δεν απορροφώνται δυστυχώ πολλέ φορέ συνοδεύονται από τέτοιε προποθέσει ώστε δεν είναι δυνατόν να απορροφηθούν τα κονδύλια αυτά. Θα πρέπει να σκεφτούμε για τον λόγο αυτό πώ θα μπορέσουμε να φτάσουμε του πραγματικού <clears throat> αποδέκτε με τον τρόπο με τον οποίο προσδιορίζουμε τα κονδύλια αυτά. Ο υποχρεωτικό χαρακτήρα, ο δεσμευτικό χαρακτήρα είναι πολύ σημαντικό από αυτή την έποψη και η πρότασή μα είναι ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις λεγόμενες επενδύσεις ε, περιοπής οι οποίες θα κατευθυνθούν προς τις περιοχές αυτές, τις μικροπεριοχές, ώστε να επιτύχουν να υπάρχει ένα ελάχιστο επίπεδο παροχών. Και αν αυτές οι περιοχές δεν, <clears throat> δεν επιτύχουν να χρησιμοποιήσουν πραγματικά αυτά τα κονδύλια, τότε τα κονδύλια πρέπει να πάνε σε άλλες περιοχές. Είναι απαραίτητο λοιπόν να υπάρξει η δυνατότητα προγραμμάτων εκπαίδευσης και ενσωμάτωσης στις περιοχές αυτές. Αν τα χρήματα αυτά λοιπόν δεν πιάνουν τόπο για να το πω έτσι, θα πρέπει να επενδυθούν σε άλλους χώρους. Η τελευταία μου παρατήρηση τώρα αφορά τις επαφές με τους φορείς των Ρώμα. Στην Ουγγαρία έχουμε ένα σύστημα βάσει του οποίου σε τοπικό, σε ενδιάμεσο και σε εθνικό επίπεδο υπάρχει ένα τέτοιο σύστημα διαλόγου Επί εθελοντικής βάσης λοιπόν μπορούν να έρθουν σε επαφή με τις αρχές η Ρώμα. Και υπάρχουν και οι εκλεγμένοι το Ρώμα. Υπάρχουν κάπου 4.800 άτομα τα οποία έχουν εκλεγεί σε τοπικό επίπεδο. Έχουν και ένα κοινοβούλιο των Ρωμά με 350 μέλη και ένα πρόεδρο. Και αυτό το όργανο, είναι και ένας εταίρος για την Ουγγρική κυβέρνηση για τα θέματα των Ρωμά. Έχουμε τη δυνατότητα αυτή λοιπόν με αυτή την αυτοδίκηση των Ρωμά να εκπροσωπούνται οι εθνικές, οι εθνοτικε μειονότητες στην Ουγγαρία. Και μια τελευταία παρατήρηση, εγώ δεν συνέδεσα ποτέ τους Ρωμά με την εγκληματικότητα, δεν μίλησα για εγκληματικότητα των Ρωμά. Εγώ νομίζω ότι αυτό δημιουργεί σε λανθασμένες εντυπώσεις και λανθασμένα συμπεράσματα κάθε ε, άτομα το οποίο έχει κάνει μια δικοπραξία έχει ένα όνομα και αυτό το όνομα είναι όνομα ανθρώπου και όχι ομάδας. Θα πρέπει πάντα να ε, μιλάμε για την εγκληματικότητα των Ρώμα, αλλά οι Ρώμα σε αυτήν την περίπτωση είναι θύματα. Πηγαίνω στην Ζηρίχη αύριο, όπου πρόκειται για την περίπτωση μιας κοπέλας που έχει έρθει από την Ουγγαρία στα 16 της και την πουλήσανε για εκπόρνευση. Είναι απαραίτητο λοιπόν στον τομέα αυτό να υπάρξει μια συνεργασία και μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών για να εμποδίσουν τέτοιου είδου εκμετάλλευση ανθρωπίνων ατόμων, ανθρωπίνων όντων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και η τελευταία μου παρατήρηση είναι σημαντικό όταν μιλάμε για την ε, συμπερίληψη και την, την ε, ενσωμάτωση να μην μιλάμε για απορρόφηση από την κύρια πολιτιστική ομάδα. Εμείς μιλάμε για να δώσουμε την ευκαιρία στους ανθρώπους αυτούς και από εκεί πέρα αυτοί θα πρέπει να αποφασίσουν ποιο κομμάτι της δικής τους κουλτούρας θα πρέπει να κρατήσουν και σε ποιο βαθμό θα δεχθούν τις ε, συνθήκες ζωής και την κουλτούρα του κράτους στο οποίο ζουν. Αυτό είναι ένα θέμα ταυτότητος, είναι μια προσωπική τους επιλογή. Πρέπει να τους δώσει κανείς ίδιες, ίσες ευκαιρίες με όλους τους άλλους σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, σε ό,τι αφορά την απασχόληση, σε ό,τι αφορά την παροχή υγειονομικής περίθαλψης την εξασφάλιση της ευμάρειά του κτλ. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Μπάλοκ. Θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της σημερινής ακρόασης. Όχι, ζητώ συγγνώμη, λέει η Πρόεδρος. Ε, βιάστηκα, θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια για να απαντήσει στις παρεμβάσεις και ερωτήσεις που έγιναν. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πολύ σύντομη, διότι βλέπω ότι ήδη έχουμε καθυστερήσει και κάποιοι πρέπει να φύγουν. Ναι, ε, δεν έχουμε ξεφύγει από το χρονοδιάγραμμα, αλλά αυτοί που θα έπρεπε να απαντήσουν έχουν ήδη φύγει. Θα, απαντήσω λοιπόν στις ερωτήσεις που τέθηκαν σε μένα. Όσον αφορά ε, το έγγραφο αυτό και γιατί ε, δεν ε, αντιμετωπίζει κάποια θέματα. Το έγγραφο αυτό ασχολείται με ένα θέμα με το οποίο ε, ασχολείται το Κοινοβούλιο εδώ και τέσσερα χρόνια. Αλλά δεν θέλουμε Ε, να είμαστε πολυαόριστοι, διότι θέλουμε να ε, σεβαστεί η Κομισιόν ε, αυτό που θα αναφέρει το Κοινοβούλιο. Το έγγραφο λοιπόν αυτό αναφέρεται σε χρηματοδότηση, νομική βάση κτλ. Οι Ρώμα μόνοι τους μπορούν να λύσουν τα θέματα που αφορούν αυτούς αποκλειστικά, τον πολιτισμό των Ρώμα, την ταυτότητα των Ρώμα κλπ. στο κέντρο της Βουδαπέστης εδώ και 40 χρόνια έχουμε ε, τραγουδιστές ε, ράπερ. Ε, η ταυτότητα των Ρώμα και η δεσμή των Ρώμα με τις πατρίδες τους έχει πληγεί πολύ από την πολιτική και των κομμουνιστών και άλλων φορέων στο θέμα αυτό τα τελευταία δεκα, ε, τις τελευταίες δεκαετίες ε, η πολιτική μας έχει βλάψει πολύ και γι' αυτό έχω συγγράψει το έγγραφο αυτό και έχω επικεντρωθεί στα θέματα που δεν είναι θέματα των Ρώμα, είναι θέματα ε, βασικών δικαιωμάτων των πολιτών της Ευρώπης. Ε, και γι' αυτό μιλάω εδώ για τη δεύτερη και τρίτη γενιά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, το δικαίωμα σε μια καλή ζωή, το δικαίωμα σε μια εκπαίδευση ποιότητα. Νομίζω ότι αυτά είναι τα σημαντικά θέματα ε, τα οποία θα πρέπει να προσέξει η Ευρωπαϊκή Ένωση και με τα οποία θα πρέπει να συμμορφωθούν τα κράτη-μέλη. Περνάμε μια δύσκολη η ιστορική περιοχή. Ε, κάποια θέματα δεν αφορούν μόνο τη μειονότητα, αφορούν και τον υπόλοιπο πληθυσμό. Υπάρχει, υπάρχουν κάποιες οικονομικές ανάγκες στις διάφορες χώρες. Ε, πολλά πράγματα λοιπόν ε, δεν έχουν τονιστεί επαρκώς τα τελευταία χρόνια και δεν θέλουμε να ασχοληθούμε τώρα με θέματα γλώσσας, ε, πολιτισμού και ταυτότητας. Πιστεύω ότι με το έγγραφο αυτό βασιζόμαστε στις εμπειρίες των ε, οργανώσεων των πολιτών που συμπαραστάθηκαν στους Ρώμα τα τελευταία 20 χρόνια. Οι κυβερνήσεις δεν έχουν συμπαρασταθεί. Πολύ συχνά οι ίδιοι οι ηγέτες τους ε, δεν ε, συμπαραστάθηκαν. Οι μη κυβερνήσει ε, δεν είχαν σκοπό το κέρδος, συμπαραστάθηκαν στους Ρώμα. Το έγγραφο αυτό βασίζεται στις δικές τους εμπειρίες και στις δικές τους προτάσεις. Το κοινοβούλιο μας είχε την τύχη επανειλημμένα να ακούσει όλες αυτές τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και νομίζω ότι σήμερα αυτός είναι ένας λόγος που εκπροσωπούνται εδώ τόσες μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Και το έγγραφο του Κοινοβουλίου ε, αλλά και της Κομισιόν ε, βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στις εμπειρίες ε, των μη κυβερνητικών οργανώσεων των Ρώμα και τις μη οργανώσεις και τις άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις. Οι εμπειρίες αυτές προέρχονται από την πραγματική ζωή, από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και από επιστημονικές έρευνες. Και δείχνουν πώς οι πολιτικές αυτές τελικά οδηγούν σε διακρίσεις. Δείχνουν πώς ε, οι ευκαιρίες ε, απασχόλησης δεν λειτουργούν στους Ρώμα. Και οι τελευταίες εξελίξεις λοιπόν είναι γνωστές στους ανθρώπους που εργάζονται με τα θέματα αυτά. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε σε διαπραγματεύσει να περάσουμε σε ένα επόμενο βήμα και με το Συμβούλιο και την Κομισιόν και ότι όλοι οι πολιτικοί φορεί θα ενωθούν ώστε να πετύχουμε κάτι νομικά δεσμευτικό, κάτι με επαρκή χρηματοδότηση και κάτι το οποίο χρειάζεται πολύ η Κομισιόν, τα κράτη-μέλη τα κράτη-μέλη να μην μπορούν να κρύψουν το θέμα των φτωχών και των ανθρώπων που χρειάζονται τη βοήθειά τους. Ευχαριστώ πολύ. I think it was very important you... Πολύ σημαντικά ήταν αυτά που μας είπατε. Και τώρα. Περνάμε στο δεύτερο τμήμα της ε, ακρόασής και για το δεύτερο αυτό τμήμα θα έχουμε τέσσερις ομιλητές. Ο κύριος Έρησης Κλούνα, ο οποίος προβλεπόταν να έρθει σήμερα, θα έρθει μόνο αύριο. Τέσσερις ήταν οι ομιλητές μας. Ο κύριος Μόρτεν Κίρομ, διευθυντής του Ευρωπαϊκού Φορέα για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα, <clears throat> ο κύριος Μπέρναρτ Ρόρκε, διεθνές διευθυντής για διεθνή έρευνα και υποστήριξη από το Ίδρυμα Ανοιχτή Κοινωνία, τον κύριο Βαλέριου Νοκάλιο, από το Κέντρο Πολιτική για του Ρώμα και τι Μειονότητε και τον κύριο Ιβάν Ιβάνοφ, Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Γραφείου Πληροφορία για του Ρώμα. Μετά από του τέσσερι αυτού ομιλητέ, επανερχόμαστε σε ερωτήσει και απαντήσει και <clears throat> συζήτηση γενικού χαρακτήρα. Πρώτα λοιπόν ζητώ από τον κύριο Κύρουμ, το Διευθυντή του Φορέα για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα, να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε να ε, μιλήσω για το πολύ επίκαιρο αυτό θέμα, ε, ειδωμένο υπό το φως των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρώπη. Όπως ε, γνωρίζετε, η Υπηρεσία Ανθρωπίνων ε, Δικαιωμάτων, ε, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ε, συλλέγει στοιχεία σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα των Ρώμα και έχουμε εξετάσει θέματα ε, απασχόλησης, εκπαίδευσης, καθώς και θέματα απλών διακρίσεων. Όλοι οι τομείς αυτοί αντιστοιχούν σε θεμελιώδη δικαιώματα ε, όπως ε, έχουν θεσπιστεί στον ε, νομικά δεσμευτικό χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα ισχυρό πλαίσιο για μια προσέγγιση βασισμένη στα δικαιώματα για να αντιμετωπίσουμε το θέμα των Ρώμα. Θα επανέλθω σε αυτό. Οι εκθέσεις που έχουμε δημοσιεύσει για τους Ρώμα συνεχίζουν να τονίζουν ότι υπάρχουν υψηλά επίπεδα διακρίσεων και ανισοτήτων. Οι Ρώμα είναι η πιο ευάλωτη ομάδα στις ε, διακρίσεις και στο ρατσιστικό έγκλημα στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύντομα λοιπόν καταρχήν να σας δώσω κάποια από τα στοιχεία από τα τις πιο πρόσφατες έρευνές μας. Ε, η έρευνα μας σχετικά με ε, τις εμπειρίες διακρίσεων ε, των ε, μικρών κοινοτήτων δείχνει ότι τουλάχιστον η μισή Ρώμα την προηγούμενη τη χρονιά πριν την εκπόνηση της έρευνας είχαν εμπειρίες διακρίσεων και μάλιστα επανειλημμένα. Οι Ρώμα είχαν ένα από τα πιο υψηλά ποσοστά ρατσιστικής βίας κατά μέσο όρο τέσσερα περιστατικά επίθεσης ή σοβαρής παρενόχλησης μέσα σε 12 μήνες. Αυτό δείχνει ότι το ρετσιστικό έγκλημα αποτελεί καθημερινή εμπειρία όλων των Ρώμα. Πέρα όμως από τις διακρίσεις ε, και την ε, ε, θυματοποίηση, οι Ρώμα αντιμετωπίζουν και δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, την εκπαίδευση και την υγεία, κάτι που οδηγεί και σε υψηλά επίπεδα ανεργίας. Όσον αφορά την ανεργία, στα 7 κράτη-μέλη που εξετάσαμε, η ανεργία μεταξύ των Ρώμα των ανδρών έφτανε το 20% κατά μέσο όρο σε, αντίθεση με, σε σύγκριση με το 7% στον γενικό πληθυσμό και στα 7 κράτη-μέλη που εξετάσαμε, τα αποτέλεσματα δείχνουν συνεχή υψηλά ποσοστά των Ρώμα ε, που να έχουν λάβει μόνο 5 χρόνια ε, βασική εκπαίδευση, σχολική εκπαίδευση στο σχολείο. Υπάρχουν ε, διαφορές ε, στα ποσοστά από χώρα σε χώρα, αλλά πάρα πολλοί είπαν ότι έχουν ε, λάβει σχολική εκπαίδευση λιγότερο από πέντε χρόνια και αν το συγκρίνουμε αυτό με τον γενικό πληθυσμό αντιστοιχούν στο 2 με 6% του γενικού πληθυσμού, ενώ μιλάμε για ποσοστό 55 με 60% μεταξύ των Ρώμα. Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα αποτελέσματα όσον αφορά την εκπαίδευση όταν κοιτάμε και τα φύλλα διότι στο γενικό πληθυσμό οι διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης είναι, η διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι πολύ μικρή. Στην περίπτωση των Ρώμα η διαφορά είναι σημαντική. Οι γυναίκες ε, λαμβάνουν περίπου το, μισό της εκπαίδευσης που λαμβάνουν ε, οι άντρες. Ε, τέλος, όσον αφορά τη στέγαση, ο μεγάλος πληθυσμός των, ε, η μεγάλη πλειοψηφία των Ρώμα δεν ταξιδεύουν και γι' αυτό χρειάζονται επαρκή ε, μόνιμη στέγαση. Ωστόσο, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα μπορούσαν να κάνουν πολύ περισσότερα, δείχνουν οι μελέτες μας. Δεν θα σας κουράσω με πολλά νούμερα, θα τα βρείτε όλα στις εκθέσεις μας. Να αναφερθώ τώρα στην κατάσταση των Ρώμα και τους ε, πιθανούς ε, δρόμους προόδου όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η κατάσταση των ε, Ρώμα αποτελεί πρόκληση για το όραμά μας της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου υπάρχει σεβασμός όλων των ανθρώπων, υπάρχει πρόσβαση των, σε δικαιώματα μη διακρίσεων. Μιλάμε για μια Ευρωπαϊκή Ένωση όπου ο κόσμος μπορεί να αισθάνεται ασφαλής. Ε, σας ανέφερα κάποιες στατιστικές. Ε, θα πρέπει να θυμόμαστε όμως ε, ότι τα νούμερα αυτά αντιπροσωπεύουν πραγματικούς ανθρώπους οι οποίοι επί χρόνια έχουν αποκλειστεί κοινωνικά εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να μην ξεχνάμε ότι την τελευταία δεκαετία ε, η πολιτική δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και η χρηματοδότηση για την ε, κοινωνική ένταξη στο Ρώμα έχει ε, δράσει ως καταλήτης ιδιαίτερα στις ε, κεντρικές ε, και ανατολικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι χώρες αυτές έχουν αντιμετωπίσει μια σειρά προκλήσεων ε, προσπαθώντας να εφαρμόσουν σχέδια δράσης για τους Ρώμα. Αυτό θα πρέπει να αναγνωριστεί και σε διοικητικό επίπεδο. Έχουν αντιμετωπίσει και πολλές προκλήσεις για την καταπολέμηση διαφόρων προκαταλήψεων. Ωστόσο, οι, τροποποίησεις, οι αλλαγές θα πρέπει να γίνουν πολύ πιο γρήγορα, οι δράσεις θα πρέπει να συντονιστούν καλύτερα, να παρακολουθούνται καλύτερα και να αξιολογούνται καλύτερα. Η η υπηρεσία μας συμμετέχει στην Task Force για τους ε, Ρώμα, την ομάδα κρούσης που ανέφερε η Vivian Redding. Πρέπει τα κράτη-μέλη να συντονίζουν και να ανταλλάσσουν ευέλτιστες πρακτικές. Αυτό σίγουρα θα είναι ωφέλιμο. Χρειάζεται όμως να υπάρχει η αίσθηση συνειδιοκτησίας μεταξύ των ε, τοπικών και εθνικών αρχών ε, και μεταξύ των ιδίων των Ρώμα. Πολλά αποτελέσματα Πολλά καλά αποτελέσματα έχουμε από τα κράτη-μέλη. Ωστόσο, οι έρευνές μας δείχνουν ότι οι δράσεις ε, που ε, αναλαμβάνονται απαιτούν πολύ περισσότερη παρακολούθηση, αξιολόγηση και φυσικά χρηματοδότηση. Ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρχει συνοχή όσον αφορά τους ε, συνδέσμους με όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και τις πολιτικές. Είναι πολύ σαφής η ανάγκη να συμπεριλαμβάνεται η πτυχή των νόμων σε όλες τις πολιτικές οι πολιτικές αυτές θα λειτουργήσουν καλύτερα οι ερευνές μας όπου, υπάρχει, ε, όπου υπάρχουν βιώσιμε πολιτικές, στι ε, στις περιπτώσεις δηλαδή όπου οι Ρώμα συμμετέχουν ήδη από τη φάση του προγραμματισμού μέχρι και την φάση της αξιολόγησης, όπως τόνισε η Λίδια Γιαρόκα στην έκθεσή της ε, σχετικά με την στρατηγική τη ε, της Ένωση για την κοινωνική ένταξη των Ρώμα, ακόμα και αν ε, θα μπορούσαμε να εξαλείψουμε τις ε, προκαταλήψεις, τις διακρίσεις, ε, ο κοινωνικός αποκλεισμός στον Ρώμα θα παρέμενε. Θα πρέπει λοιπόν να εφαρμόσουμε αντιρρεσιστικά μέτρα παράλληλα με τα μέτρα κοινωνικής ένταξης. Αυτά θα πρέπει να τα συνδέσουμε και με δράσεις που να βελτιώνουν τις κοινωνικές συνθήκες των ε, Ρώμα που στερώνονται βασικών αγαθών και που είναι κοινωνικά αποκλεισμένοι. Ε, το ίδιο ισχύει και για τους ε, και για ανθρώπους που δεν είναι Ρώμα, που μένουν όμως μαζί τους στις ίδιες κοινότητες. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι συχνά οι δράσεις για την ένταξη των Ρώμα αντιμετωπίζονται με εχθρότητα από μη Ρώμα, όταν έχουν σχεδιαστεί με τρόπο που να αποκλείουν τους μη Ρώμα εντός της ιδίας τοπικής κοινωνίας. Γι' αυτό οι δράσεις ένταξης θα πρέπει πάντα να αποτελούν μέρος μιας ε, μέτρων γενικότερης ε, οικοδόμησης των κοινοτήτων και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν και τους Ρώμα και τους μη Ρώμα. Αυτή η προσέγγιση έχει θετηθεί από την Στρατηγική Ευρώπη 2020 ε, στην πρωτοβουλία πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της φτώχειας που στόχο έχει να πετύχει εδαφική συνοχή και να πετύχει και σεβασμό των θεμελιωτών δικαιωμάτων όλων ε, όσων ε, ζουν υπό συνθήκε φτώχεια και κοινωνικού αποκλεισμού. Η, Ευρω... η Στρατηγική Ευρώπη 2020 τονίζει και την σημασία των ε, τοπικών και περιφερειακών αρχών για την εξέβρεση βιώσιμων λύσεων. Η Στρατηγική Ευρώπη 2020 μπορεί να αποτελέσει καλή ευκαιρία και να ε, εφαρμόσει και κάποιους, κάποιους επιμέρους στόχους όπως είναι η ε, κοινωνική ένταξη των Ρώμα και μη Ρώμα. Ε, το να έχουμε επιμέρους στόχους ε, μας βοηθάει να έχουμε καλό μέτρο του αντικτύπου των διαφόρων πολιτικών. Μια ε, προσέγγιση που να βασίζεται στα θεμελιώδη δικαιώματα μπορεί να αποτελέσει στόχο που να ασχολείται με του Ρώμα αλλά και τον γενικό πληθυσμό σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές. Να κλείσω λέγοντα ότι βασίζω, ε, με βάση τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει και αναλύσει, είναι σαφές ότι το θέμα της ένταξης στο Ρώμα μπορεί να αντιμετωπιστεί καλύτερα με μια ολιστική προσέγγιση, να έχουμε καταρχήν μία ε, εγκάρσια προσέγγιση ε, από τη βάση προς τα πάνω που να συνδέει ε, το τοπικό, το εθνικό και το ευρωπαϊκό επίπεδο. Χρειαζόμαστε επίσης μια οριζόντια προσέγγιση που να συνδέει τις δράσεις στους κυρίους τομείς παρέμβασης όπως είναι η στέγαση, η εκπαίδευση και η υγεία. Τέλος, πιστεύω ότι δύο θέματα θα είναι βασικά στις περαιτέρω δράσεις. Καταρχήν, η πραγματική συμμετοχή των Ρώμα και των μη Ρώμα στον σχεδιασμό και την ε, υλοποίηση των δράσεων, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο. Αυτό θα διασφαλίσει οι δράσεις να καλύπτουν τις πραγματικές τους ανάγκες και όχι αυτό που θεωρούν άλλοι ότι είναι οι ανάγκες τους. Αυτό θα οδηγήσει σε πολύ καλύτερη αποδοχή των πολιτικών και των μέτρων από τους Ρώμα, όπως έχουν δείξει οι έρευνές μας στον τομέα της στέγασης, για παράδειγμα. Και από την άλλη μεριά, όπως είπε πρόσφατα το Ινστιτούτο Ανοιχτής Κοινωνίας, αν δεν υπάρχουν δεδομένα δεν υπάρχει πρόοδος. Δεν μπορούν να σχεδιαστούν δράσεις, ούτε μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο παρακολούθηση και αξιολόγηση αν δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία. Εάν δηλαδή δεν γνωρίζουμε ποια είναι πραγματικά η κατάσταση. Και μπορώ να σα διαβεβαιώσω ότι ε, η Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα συνεχίσει την ε, ει εργασία μα, την αναλυτική εργασία μα στον τομέα αυτών για να εργαστούμε με στόχο πολύ υψηλότερο επίπεδο προστασία των δικαιωμάτων των Ρώμα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Κύρουμ. Δίνω το λόγο στον κύριο Μπέρναντ Ρόρκ από το Ίδρυμα Ανοιχτής Κοινωνίας. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την ευκαιρία που μου δίνετε να λάβω το λόγο ενώπιον της ακροάσεως σας εδώ σήμερα. Πριν από πολλά χρόνια, θυμάμαι, κάποιοι από εμά ζητήσαμε μια πλήρη πανευρωπαϊκή στρατηγική για του Ρωμά. Μας είπανε, δεν γίνεται αυτό, είναι αδιανόητο, είναι εκτός των αρμοδίων τίτων της Ευρωπαϊκής Ένωση και της ε, Κομισιόν. Τώρα, μετά από την δεύτερη διάσκεψη κορυφής για του Ρώμα την προηγούμενη, τον προηγούμενο Απρίλιο, η ανακοίνωση τη Κομισιόν δείχνει το δρόμο, τονίζει τη σημασία μια συνεκτικής πολιτικής η οποία είναι αναλογική στην κλίμακα του προβλήματος που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. εμείς επιμένουμε ότι η κύρια ευθύνη για την ασφάλεια και την ακαιρεότητα των πολιτών μιας χώρας για την στέγαση, για την υγεία και την ευμάρειά τους ανήκει στα εθνικά κράτη. Αλλά τα έχουν κάνει τόσο θάλασσα τα εθνικά κράτη, ώστε να αφήνουν να εννοηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να έχει ένα σημαντικό ρόλο να παίξει στον τομέα αυτό. Η κυρία Ρέντινγκ είναι έτοιμη να διαμεσολαβήσει μεταξύ των κρατών μελών, να καταγράψει την ε, πρόοδο η οποία έχει επιτευχθεί, την έλλειψη τη πρόοδου. Αυτό λοιπόν πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Χρειάζεται να υπάρξει μια στοχοθεσία για του Ρώμα, όχι αποκλειστικά όμω μόνο για αυτού, ώστε τα αναπτυξιακά ταμεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορούν να καλύψουν, παραδείγματο χάρη, τη στέγαση των Ρώμα αυτή η στοχοθεσία πρέπει να είναι στοχευμένη στους Ρωμά χωρίς να είναι αποκλειστική, θα πρέπει να διατρέχει όλη την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε αυτές οι παρεμβάσεις να βοηθήσουν πάρα πολλούς Ρωμά να βγουν από τις τρόγλες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να περάσει το επίπεδο της διαμεσολάβησης, θα πρέπει να δημιουργήσει μέτρα βαθμολόγησης και δείκτες που να καταγράφουν την πρόοδο της ε, κατάστασης στο Ρώμα. Αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί, δεν πρέπει απλώς να φύγουμε από την αίθουσα με την εντύπωση ότι κάτι έχουμε επιτύχει για κάποια ασαφή μορφή <clears throat> συνένεσης μεταξύ μας. Ο κύριος φόρος, φόβος μου είναι ότι οι προσπάθειές μας, οι συστάσεις μας, οι διαβουλεύσεις μας δεν θα οδηγήσουν τίποτα σε τίποτα άλλο παρά ένα ανώδυνο, σε ένα ανώδυνο ανακοινωθέν τον επόμενο Απρίλιο. Που θα γίνεται καλή την πίστη, θα είναι έμπλεος καλών προθέσεων, αλλά δεν θα έχει κανένα πραγματικό περιεχόμενο. Ελπίζω να διαψευστώ. Γνωρίζω ότι υπάρχουν όρια στο τι μπορεί να επιτύχει η Κομισιόν και εκτιμώ ιδιαίτερα τις προσπάθειες του αφοσιωμένου προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα αυτά που έχουν κάνει για να προωθήσουν την ενσωμάτωση των Ρωμά. Χρειαζόμαστε όμως μια νέα εκκίνηση, μια ριζικά διαφορετική εκκίνηση. Το ανακοινωθέν του περασμένου Απριλίου θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο η ετήσια έκθεση παρακολούθησης της Κομισιόν για να επιταχύνει την ε, πρόοδο δείχνει τις τεράστιες αποτυχίες που είχαμε σε πάρα πολλούς τομείς. Αν θέλουμε στην πλατφόρμα για τους Ρωμά να ξεπεράσουμε <clears throat> τις απλές, ε, τα απλά ευχολόγια και τις καλές προθέσεις, θα πρέπει να θέσουμε σαφείς στόχους και να έχουμε μια αυστηρή παρακολούθηση το πώς χρησιμοποιούνται τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Η τωρινή Task Force έχει μια ζωή μόνο έξι μηνών. Είμαστε τυχεροί που υπάρχει μια, βρισκόμαστε σε μια εποχή που η Τρόικα η Ισπανικής, Βελγικής και Ουγγρική Προεδρία έχει θέσει το ζήτημα το Ρωμά στο κέντρο των ενδιαφερόντων της και υποστηρίζει την ανάγκη μιας συνέχεια της στρατηγικής για τους Ρωμά. Τι θα γίνει όμως μετά την Ουγγρική Προεδρία στην πλατφόρμα για τους Ρωμά. Πρέπει να υπάρξει μια μόνιμη task force η οποία θα συνεχίσει την πορεία αυτή η οποία ξεκινήσει. Πρέπει να υπάρχει μια βιώσιμη αλλαγή γιατί η τωρινή κατάσταση δεν είναι βιώσιμη. Για να το πω όμα, όσο αντιμετωπίζουν αποκλεισμό και αποξένωση οι Ρωμά στι χώρε του, θα εξακολουθήσουν να μεταναστεύονται. Να μεταναστεύουν. Και η μετανάστευση και όχι τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής των Ευρωπαίων πολιτικών. Το να αντιμετωπίσουμε τους κύριους λόγους, όπως είπε η Επίτροπος Ρωμά, που οδηγούν τους Ρωμά στο να μετακινούνται από τις χώρες τους και να έρχονται στην Ευρώπη, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο, γιατί χωρίς την αντιμετώπιση αυτή μπορεί η ατζέντα να καθορίζεται από λαϊκιστές και ακροδεξιούς ρατσιστές. Χωρίς λοιπόν μια σωστή αντιμετώπιση δεν μπορούμε να έχουμε μια συνεκτική πολιτική. Αν παραμείνουμε, όπως είπε η κυρία Ρέντινγκ, κοινότη αξιών και θεμελιωδών δικαιωμάτων. Θα πρέπει να είμαστε επάγρυπνοι ενώπιον όλων αυτών οι οποίοι ουσιαστικά ε, είναι έτοιμοι να καταπατήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να περιγελάσουν τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα από τα βασικά προβλήματα καταρχήν είναι ο διαχωρισμός στα σχολεία και η πρακτική να θεωρούνται τα παιδιά το Ρωμά ότι είναι πνευματικά υπολοιπόμενα και να τα στέλνουν σε ειδικά σχολεία. Είναι κάτι το ανησυχητικό ότι τα κράτη-μέλη εξακολουθούν να ακολουθούν αυτή την πρακτική παραβιάζοντας τις αποφάσεις που έλαβε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εναντίον της Τσεχικής Δημοκρατίας πριν από τρία χρόνια. Οι έρευνες του Ταμείου για την εκπαίδευση των Ρωμά δείχνουν ότι αυτές οι πρακτικές συνεχίζονται σε χώρες όπως η Σλοβακία. Ο αριθμό των παιδιών που πήγαν σε ειδικά σχολεία αυξάνεται. Αυτές οι πρακτικές αντιβαίνουν σε οποιαδήποτε ένταξη έννοια ένταξη των Ρωμά. Θα πρέπει όλα τα κράτη-μέλη να κάνουν προσπάθειες να σταματήσουν αυτό το apartheid κατά των παιδιών. Πρέπει ήδη από τα προσχολικά προγράμματα να εξασφαλίσουμε ότι τα παιδιά των Ρωμά είναι έτοιμα για το σχολείο και ότι υπάρχει ένα ενσωματωμένο περιβάλλον μάθηση όπου τα παιδιά των Ρωμά δεν αντιμετωπίσουν διάκριση και ότι οι διδάσκαλοι του είναι έτοιμοι να αποδεχτούν και να δουλέψουν με την πολυμορφία. Η στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δώσει έμφαση στην ευμάρεια των παιδιών των Ρωμά. Αυτό είναι στην καρδιά της ανθρώπινης ανάπτυξης. Όταν μειώνεται διογραφικά ο πληθυσμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ρωμά είναι το ταχύτερα αναπτυσσόμενο δημογραφικά τμήμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέραν τη ηθική επιταγή, η ευρωπαϊκή κοινωνία δεν μπορεί να δεχτεί άλλη μια χαμένη γενιά αποκλεισμένων από την κοινωνία νεαρών Ρωμά έχουμε προειδοποιήσει ότι μπορούμε να έχουμε μια ευρωκεντρική και μειοπική αντιμετώπιση. Πρέπει να έχουμε μια πλήρη στρατηγική για τη συμπερίληψη των Ρωμά και μια τέτοια στρατηγική για να είναι πραγματικά πανευρωπαϊκή πρέπει να λάβει υπόψη και τα Δυτικά Βαλκάνια. Θεωρούμε ότι επίση χρειάζεται πολύ περισσότερη προσπάθεια για να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχή στην κοινότητα των Ρωμά. Λέμε πολύ συχνά ότι η ένταξη είναι μια αμφίδρομη διαδικασία. Αλλά εάν η ουσία της συμμετοχή στο Ρωμά δεν εξασφαλιστεί, θα μείνει καινογραμμά όλη αυτή η διαδικασία. Χωρίς διαβούλευση, χωρίς διάλογο για να κατανοήσει κανείς τις επιθυμίες των κοινοτήτων αυτών και, τα, και τις προσδοκίες τους, χωρίς να υπάρχει συμμετοχή τους στην ανάπτυξη πολιτικών ενσωμάτωση, οι μελλοντικέ προσπάθειες θα είναι τόσο αναποτελεσματικέ όσο και οι προηγούμενε μια στρατηγική πλαισίου θα πρέπει να προωθήσει την ενεργή συμμετοχή των Ρώμα ως πολιτών και όχι μονάχα ως αποδεκτών, παθητικών αποδεκτών. Μόνο χάρη στους ακτιβιστές των Ρωμά τα τελευταία δέκα και παραπάνω χρόνια υπήρξε αναγνώριση των ε, Ρωμά, του προβλήματος των Ρωμά. Μη κυβερνητικοί φορεί οι οποίοι συνδέονται με τι τοπικέ κοινότητε έχουν παίξει επίση το ρόλο των υπερμάχων των δικαιωμάτων των Ρωμά και έχουν παίξει σημαντικό ρόλο. Αλλά για εκατομμύρια Ρωμά όλα αυτά τα οποία λέγονται για την κοινωνία των πολιτών δεν σημαίνουν τίποτα άλλο, γιατί δεν έχουν καν έρθει σε επαφή με τους ακτιβιστές των ίδιων των Ρωμά. Σε σχέση με το μέγεθος του πληθυσμού, η κοινωνία των πολιτών είναι πάρα πολύ ισχνή ακόμα. Χρειάζεται να δώσουμε προτεραιότητα σε μια, μια ισχυ, ισχυροποίηση του τομέα της κοινωνίας των πολιτών και υπάρχει ανάγκη για όλους τους εμπλεκομένους να συντονίσουν τη δράση τους και να έχουν μια συνεκτική δράση για να δώσουν τις απαραίτητες δεξιότητες στους φορείς των Ρώμα. Ξεκινώντας από το μηδέν σε πόλεις και σε χωριά όπου δεν υπάρχει καθόλου αυτή η δυνατότητα. Πρέπει να εξασφαλίσουμε επίση και την ισότητα των φύλων και τη συμμετοχή των γυναικών Ρωμά για να αντιμετωπίσουν την πολλαπλή διάκριση που αντιμετωπίζονται. Πρέπει και αυτό να είναι στην καρδιά όλων των παρεμβάσεων. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα στερεότυπα και τι προκαταλήψει, να αντιμετωπίσουμε το ρατσιστικό και ξενοφοβικό λόγο σε πολιτικό επίπεδο και την ε, ε παρότρινση σε σε βία και μίσος και την παρέμβαση των ακροδεξιών κομμάτων που στρέφονται εναντίον των Ρώμα. Χρειαζόμαστε σωστή ευκυβερνησία στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντιμετωπίσουμε τις ρατσιστικές αυτές αντιμετωπίσεις και να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα δημόσια όργανα θα λαμβάνουν υπόψη πλήρω την ιδέα της μη διάξης. Δεν χρειαζόμαστε σε επίπεδο δημοσίων εκστρατιών και άλλες πρωτοβουλίες οι οποίες είναι μεγαλώσιμε μεν αλλά χωρίς αποτελέσματα. Πρέπει να προχωρήσουμε πέραν αυτών και επέκεινα αυτών και να ξεπεράσουμε απλώ τι πόλεις. Πρέπει να πάμε στις κομοπόλεις και στα χωριά όπου οι εντάσει με του Ρωμά είναι πολύ μεγαλύτερε. Θα πρέπει να συμπεριληφθούν λοιπόν σε όλα αυτά και οι μειονοτικοί και οι πλειοψηφικοί πολιτισμοί. Δεν θα πρέπει να κάνουμε προσπάθειες οι οποίες θα γίνουν σήμερα και θα χαθούν αύριο. Θα πρέπει να αφήσουμε κάποιο αποτέλεσμα. Και θα πρέπει να προωθήσουμε και τον κοινωνικό διάλογο. Το γεγονός ότι οι κοινότητε στο Ρωμά, οι οποίες χρειάζονται περισσότερα χρήματα και βοήθεια, δεν έχουν τη δυνατότητα να πάρουν χρηματοδότηση, να έχουν πρόσβαση, οδήγησε το Ίδρυμα Σόρο ανοιχτή Κοινωνίας να δημιουργήσει μια σειρά από προγράμματα τεχνικής ε, αρρωγής, υποστήριξης, παρακολούθησης, χρηματοδότησης και υποστήριξης σε διάφορα επίπεδα. Ελπίζουμε ότι αυτές οι υποστηρίξεις θα βοηθήσουν να υπάρχει στοχοθεσία, όχι αποκλειστική όμως, και επίσης με ένα συνδυασμό πολιτικών και χρηματοοικονομικών κινήτρων να φέρουν τους Ρωμά από το περιθώριο στο κέντρο της, του πολιτικού γίγνεσθε. έχουμε κάποια διδάγματα που μπορούμε να αντλήσουμε από την τελευταία δεκαετία προσπαθειών για την ενσωμάτωση των Ρωμά. Παρά τις αποτυχίες έχουμε μία, πιστεύω, ένα βασικό πλαίσιο. Η δεκαετία αυτή μας έδωσε ένα πλαίσιο τακτικής ανταλλαγής απόψεων και έχει δεσμεύσει τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κλείσουν το χάσμα σε στέγαση, απασχόληση, εκπαίδευση. Έδωσε τη δυνατότητα μεγαλύτερου συντονισμού και διαλόγου με έναν τρόπο που δεν τον επέτυχε ποτέ η ανοιχτή μέθοδος συνεργασίας δημιουργία και ένα πλαίσιο διαλόγου και ανταλλαγών απόψεων για τα κράτη-μέλη και για τις χώρες οι οποίες είναι όμορες τη Ευρωπαϊκής Ένωση και μπορούν να συμμετάσχουν πλήρως. Και συνενώνει τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και τους θεσμικούς φορείς για να μπορέσουν να φτάσουν σε συνεκτικές πολιτικές συμπερίληψεις. Από αρνητική έποψη, οι προσπάθειες αυτές έχουν προσκρούσει σε έλλειψη πολιτικής θέλησης, σε έλλειψη σαφών στόχων σε πολιτικό επίπεδο, έλλειψη σαφών δεδομένων, έλλειψη ικανότητα σε δημοτικό και τοπικό επίπεδο και απροθυμία να αντιμετωπιστεί καν το θέμα του αποκλεισμού και της διακρίσης, των διακρίσεων και τέλος της ε, έλλειψης ικανότητας να απορροφηθούν πόροι όπως αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Αυτό το οποίο χρειάζεται λοιπόν να γίνει οι χώρε οι οποίε έχουν συμμετάσχει την τελευταία δεκαετία έχουν ζητήσει από την Κομισιόν να υποστηρίξει τι προσπάθειέ του, να συν... τονίσει τι προσπάθειέ του, να εκπονήσει μια κοινή στρατηγική η οποία θα έχει και τρόπο να καταμετρά την πρόοδο. Οι εθνικέ κυβερνήσει συζητήσαν στο τέλο δεκαετίας και την παρέμβαση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει αυτή να ακολουθήσει το πνεύμα αυτό της δεκαετίας και να ενισχύσει όλες αυτές τις προσπάθειες και να εξασφαλίσει τη συνέχεια της δεκαετίας και αυτό περιλαμβάνει και τα διδάγματα από την αποτυχία της δεκαετίας που θα είναι η πρώτη ύλη για μια νέα στρατηγική ένταξης. Θα πρέπει να ξεπεράσουμε αυτή τη δεκαετία άτυπου apartheid. Χρειαζόμαστε ένα οδικό χάρτη ενσωμάτωσης που μας οδηγήσει προς το μέλλον, γιατί το παρόν για πάρα πολλούς ανθρώπους, πάρα πολλούς πολίτες της μεγαλύτερης αθνοτικής μειονότητας Ευρώπης, το παρόν είναι πολύ ζωφερό και πρέπει να μπορούν να ταινιστούν στο μέλλον. Ε, interesting. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε. Θα δώσω τώρα το λόγο. Πρέπει να συνεχίσουμε στον κύριο Βαλεριού Νικολάε. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να χρησιμοποιήσω μια παρουσίαση PowerPoint. Θα ήθελα όμως πρώτα κάτι να τονίσω κάτι που είπε ο κύριος Βαγγελίου, το οποίο θα πρέπει να πάρουμε πολύ σοβαρά. Θα πρέπει να συγκεντρώσουμε την εμπειρία που υπάρχει. Αν έχουμε προσφορά από κάποια, κάποιον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης να κάνουμε περισσότερο, θα πρέπει να το πάρουμε στα σοβαρά, διότι πιο σημαντικό είναι οι άνθρωποι που έχουν την πρακτική πείρα να κάνουν πράγματα. Εμείς μπορούμε να συζητάμε επί πολλή ώρα, αλλά τελικά οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν τη μεγαλύτερη σημασία. Θα έπρεπε να λειτουργήσει η ηλεκτρονική παρουσίαση, δεν λειτουργεί. Θα ε, σας κάνω την ομιλία μου λοιπόν χωρίς τις διαφάνειες. Ε, εκπονήσαμε ένα έγγραφο το οποίο λέγεται το αποτελεσματικό πλαίσιο για τις εθνικές στρατηγικές. Έχει σταλεί στην Κομισιόν και στα κράτη-μέλη. Έχει σταλεί και σε ευρωβουλευτές. Αναφέρεται στην ε, κατανομή καθηκόντων και ε, στην ε, συμμετοχή των ενδιαφερομένων. Αυτό είναι το πρώτο μας έπιμα. Όταν μιλάμε για την κοινωνική ένταξη των Ρώμα, θα πρέπει να σταματήσει το παιχνίδι ανάμεσα στους διάφορους φορείς. Κάποιοι μηχανισμοί χρειάζονται για να αντιμετωπιστούν τα πολύ δύσκολα θέματα. Δυστυχώς ε, ούτε η Task Force ούτε οι πλατφόρμες ε, είναι αρκετά ισχυρά προς το παρόν. Προτού να προχωρήσουμε σε λεπτομέρειες, είχα στην παρουσίασή μου Ε, βιντεάκι με πολύ καλέ εικόνε από με διάφορα μέρη στη Ρουμανία. Ήταν πολύ καλό το παράδειγμα αυτό. Το άλλο παράδειγμα που θα χρησιμοποιήσω τώρα είναι το αποτέλεσμα ενό ανθρώπου που λέγεται Μίτου Τζοζέσκου που θεωρείται Ρουμάνος, είναι πολύ πλούσιος, είναι πολύ καλά ενταγμένος στην κοινωνία της Ρουμανίας, έχει μια πολύ καλή επιχείρηση. Πήγε στη Γερμανία, στο αεροδρόμιο του Μονάχου είχε κάνει κράτηση για ε, ένα αυτοκίνητο πολυτελείας. Ε, πολύ καλή η, η πιστοτική του κάρτα, οπότε το απάντησαν ότι ναι, έχετε την, ε, σας έχουμε κάνει την κράτηση. Όταν πήγε στο Μόναχο, η κυρία στο κατάστημα πρόσεξε ότι είναι αρκετά μελαχρινός ο κύριος και είπε ότι δεν, θεώρησε ότι δεν μπορούν να νοικιάσουν στον άνθρωπο αυτόν αυτοκίνητο, και αυτό ήταν. Του είπανε ότι δεν μπορούμε να ε, νοικιάσουμε οχήματα σε Ρωμάνους πολίτες διότι τα κλέβουν και περνάνε τα σύνορα. Το πρόβλημα ήταν λοιπόν ότι το χρώμα του δέρματός του δεν αντιστοιχούσε στην, κάρτα, στην πιστοτική του κάρτα. Ο κύριος Τζοζέσκου είχε το χρήμα, το χρόνο και ε, τη διάθεση να ασχοληθεί με την υπόθεση. Αυτό δεν ισχύει για τους περισσότερους Ρώμα. Λοιπόν, μείνει την εταιρεία η Eurocar αντί να ε, απολογηθεί, ε, έστειλε ένα μάλλον ε, αγενές γράμμα, στο οποίο έλεγαν ότι, μπορούν, ότι η επιχείρηση μπορεί να αρνείται τις υπηρεσίες της προς τους πολίτες της Ανατολικής Ευρώπης λόγω των εμπειριών που είχαν στο παρελθόν. Αυτό λοιπόν μπορεί να αντιμετωπίσει ένας Ευρωπαίος πολίτης. Φανταστείτε ο Κόλιν Πάουελ να πάει στο Μόναχο και να μην τον αφήσουν να νοικιάσει αυτοκίνητο πολυτελεία, διότι η κοπέλα θα του πει ότι «Α, κοιτάξτε, οι μαύροι ε, στη Νέα Υόρκη από όπου προέρχεστε εσείς είναι γνωστοί για το ότι κλέβουν αυτοκίνητα». Ε, αυτό θα ήταν τελείως απαράδεκτο. Και αυτό θα αποτελούσε το τέλος της Eurocar. Στη συγκεκριμένη περίπτωση κανένα δεν αντέδρασε και είμαι περίεργος να δω εάν το Κοινοβούλιο, η Κομισιόν ε, ή κάποιος άλλος θα θέλει να στείλει επιστολή προς την Eurocar. Διαπιστώσαμε ότι κανένας από αυτούς τους φορείς ε, είχε τη διάθεση να κάνει κάτι. Ε, θα σας σταλώ, αν ενδιαφέρεστε, όλα τα απαραίτητα έγγραφα, αν θέλετε να απαντήσετε. Σήμερα θα επικεντρώσω την ομιλία μου σε θέματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, τα οποία όμως αγνοούνται. Το βασικό μου επιχείρημα είναι ότι οι διακρίσεις εις βάρος των ε, ε, Ρώμα ε, κάνουν αδύνατη, καθιστούν αδύνατη τον, καθιστούν αδύνατη την κοινωνική ένταξη. Ακόμα και κάποιος καλά εκπαιδευμένος Ρώμα δεν θα λάβει θέση απασχόλησης, στέγαση και οτιδήποτε άλλο. Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι αποτέλεσμα η 20 αποφυγής ευθυνών ε, καθώς και ανικανότητας ε, και έλλειψης ε, εμπειριών. Δεν έχουμε αρκετές εμπειρίες ώστε να γνωρίζουμε πώς, μπορούν, πώς μπορεί να λειτουργήσει το να διευρύνουμε προγράμματα, σε, να κάνουμε προγράμματα μεγαλύτερα, να τα ξέρουμε σε μέγεθος. Ε, οι διακρίσεις ε, εις βάρος ε, των Ρώμα σπρώχνει κάποιους ανθρώπους στο περιθώριο και τους κάνει πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Ο πληθυσμός των Ρώμα είναι πολύ ποικιλόμορφος και φαίνεται ότι ακόμα δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Ακόμα δημιουργούμε όμοιες πολιτικές για όλους τους Ρώμα. Οι πολιτικές που επικεντρώνονται τους ε, Ρώμα, αγνοούν το ε, γεγονός αυτό και ε, καταλήγουν σε μηδενικά αποτελέσματα. Συνεχίζουμε μία παράδοξη προσέγγιση. Αγνοούμε, για παράδειγμα, τις μικτές οικογένειες οι οποίες έχουν τεράστιο δυναμικό όσον αφορά την κοινωνική ένταξη. Ούτε ένα έγγραφο δεν είδα που να μιλά για το θέμα αυτό. Είμαι πεπισμένο ότι η πλειοψηφία των Ρώμα στο, στη Ρουμανία ε, έχουν ε, μεικτή προέλευση. Ε, η αντιμετώπιση απέναντι στους Ρώμα είναι μάλλον απεικιοκρατική. Χρειαζόμαστε μη κυβερνητικές οργανώσεις ε, που να ασχολούνται με την κοινωνική ένταξη, που να ασχοληθούν και με την κοινωνική ένταξη των Ρώμα. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που κάνει η κυρία Ρέντινγκ, αλλά ε, η νομιμότητά της ε, αγγίζει το μηδέν. Εάν δεν έχει κάποιον ε, στο γραφείο της ε, που να προέρχεται από τους Ρώμα, δεν ε, μπορεί να λέει ό,τι θέλει για τους Ρώμα, δεν θα έχει καμία νομιμότητα. θέλουμε να αποφύγουμε τις υπερβολικές εκθέσεις καθώς και τα ψέματα. Ε, αυτό όμως είναι η πραγματικότητα. Επικεντρωνόμαστε υπερβολικά στα θετικά αποτελέσματα ε, και τα προβάλλουμε επειδή έχουμε πληρώσει για τα έργα αυτά. Τι θα πρέπει να κάνουμε. Θα πρέπει να αλλάξουμε τις ε, αρνητικές, την αρνητική αντιμετώπιση και θα πρέπει εντός των κοινοτήτων των Ρώμα να προωθήσουμε ε, την ε, ενεργό πολιτική ζωή. Υπάρχει τεράστιο δυναμικό ε, προόδου. Χρειαζόμαστε εθνικούς εμπειρογνώμονες για τους Ρώμα και σχέδια ανθρωπίνου δυναμικού. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στατιστικά παραμένουν ε, αυτά που ε, αποκλείουν περισσότερο τους Ρώμα όσον αφορά την απασχόληση. Οι βασικές ε, ευθύνε θα πρέπει να μείνουν στα χέρια των κρατών μελών. Χρειαζόμαστε εθνικές στρατηγικές για την κοινωνική ένταξη στο Ρώμα που να βασίζονται στα διαφορετικά ταμεία και να συμπληρώνονται με πόρους και από τα, τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Χρειάζονται εδώ πέρα benchmarks, όρια αναφοράς. Χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για να, για αντιμετωπίσουμε το θέμα. Το να απελάβουμε τους ε, Ρώμα, το να τους απειλούμε με πολιτική δράση και να χρησιμοποιούμε ρατσιστική ρητορική είναι ε, ε, πολύ άκομψος τρόπος να ασχολούμαστε με το θέμα. Θα πρέπει να σχεδιαστεί η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των πολιτικών. για να βελτιωθεί η απορρόφηση των ε, πόρων ε, στην ε, Ρουμανία. Πολλοί πιστεύουν ότι θα πρέπει να υπάρχουν αρμόδιες αρχές. Κατά τη γνώμη μου είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να σκεφτούμε την κοινωνική ένταξη των Ρώμαν, να δημιουργήσουμε ένα νέο μηχανισμό για κάτι τέτοιο. Επίσης υπάρχει η ευθύνη των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων θα πρέπει να απαιτούν πραγματικές, πρακτικές εθνικές στρατηγικές με σαφείς γραμμές προϋπολογισμού, με σαφή χρηματοδότηση. Θα πρέπει οι Ρώμα να μην συμπεριληφθούν μόνο στην ε, πλατφόρμα κατά της φτώχειας Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που είναι η ασθενέστερη από τις ε, σχετικές πρωτοβουλίες. Υπάρχουν άλλες δύο πολύ πιο ισχυρές πλατφόρμες στις οποίες θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριληφθούν οι Ρώμα. Αυτή τη στιγμή η στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση 2020 δεν λέει ούτε λέξη για τους Ρώμα. Επίσης θα πρέπει να συνεχίσουμε με βάση τα βήματα που έχουν γίνει στα τελευταία χρόνια. Μετά την ε, Ουγγρική ε, Προεδρία θα έχουμε τρεις προεδρίες που δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για θέματα των Ρώμα. Εάν ε, αφήσουμε να ξεχαστούν τα καλά βήματα αυτά, δεν θα έχουμε πετύχει τίποτα. Τέλος, ε, μηχανισμοί. Χρειαζόμαστε ε, σχετικούς ε, μηχανισμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι άτοπους, το, άτυπους, συγγνώμη. Το, το Task η ομάδα κρούσης, είναι ένας τέτοιος άτυπος μηχανισμός. Η πλατφόρμα για τους Ρώμα συναντιέται δύο φορές το χρόνο, κάτι που δεν λειτουργεί πολύ καλά αυτή τη στιγμή. Χρειάζεται σημαντική βελτίωση εάν θέλουμε να λύσουμε τα θέματα αυτά. και θα πρέπει να ε, φροντίσουμε να έχουμε πολύ καλύτερους και πιο συμμετοχικούς ε, μηχανισμούς ε, διαβούλευσης από ό,τι έχουμε αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα χωρίς τους Ρώμα, εάν θέλουμε να πετύχουμε την κοινωνική τους ένταξη. Δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς, μπορείτε να το κάνετε εσείς μόνοι σας. Η κοινωνική ένταξη έχει να κάνει με τη συμμετοχή. Αυτή τη στιγμή κάποιοι από εμά βρίσκονται σε θέσεις λήψης αποφάσεων που δεν είναι Ρώμα και υπάρχει από την πλευρά των Ρώμα η προσδοκία να βελτιωθεί η κατάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, ο κύριος Ιβάν Ιβανόφ, ο οποίος είναι ο Διευθυντής του Γραφείου Πληροφοριών ε, της, του Ευρωπαϊκού Γραφείου Πληροφοριών στο Ρωμά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να συνεχίσω με την κυρία Γιαρόκα. Είσαστε η μόνη Ρωμά στο Κοινοβούλιο και έχετε πετύχει τόσο πολλά. Φανταστείτε αν υπήρχαν άλλοι πέντε ή δέκα. Θα είχαν προχωρήσει πολύ τα πράγματα ως τελευταίος ομιλητής. Ως τελευταίος ομιλητής κινδυνεύω να επαναλάβω πολλά από αυτά τα οποία ελέγχθησαν προηγουμένως. Θα προσπαθήσω όμως να αντιμετωπίσω θετικά αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Όπως είπε ο Μπερνάρ, πριν από 5-6 χρόνια δεν υπήρχε περίπτωση να μιλήσει κανείς καν για το θέμα μιας στρατηγικής, μιας πολιτικής, οτιδήποτε, που να είναι ειδική για τους Ρωμά. Τα πράγματα όμως προχωρούν. Πριν από 5-6 χρόνια, πολλοί κόσμος, και μιλάω περισσότερο για τις εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές, για την κοινωνία των πολιτών κτλ, μιλούσαν για προβλήματα. Εμείς είμαστε ακόμα στη φάση της ε, ανείχνευσης και του εντοπισμού των προβλημάτων. Τώρα μιλάμε για το τι πρέπει να γίνει. Δεν μας λέει όμως κανένας για το πώς θα πρέπει να γίνει η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Η θέση του δικού μας δικτύου είναι ότι η τελική χρησιμότητα αυτής της στρατηγικής είναι να υπάρξει μια εφαρμογή μέτρων που θα φέρει πραγματική αλλαγή στις κοινότητες στο Ρωμά ο στόχος μιας νέας στρατηγική που έχει να κάνει με του Ρωμά θα πρέπει να εξασφαλίσει πληρή και αποτελεσματική ισότητα μεταξύ Ρώμα και μη Ρώμα. Ο στόχος είναι λοιπόν να εξασφαλιστεί πλήρω η πολιτική ισότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωσης. Γιατί η Ρωμά είναι μία από τις πιο περιθωριοποιημένε ομάδες στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και επομένω μπορούν να ωφεληθούν περισσότερο από αυτή την πολιτική ισότητας τα θέματα των Ρωμά τώρα μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο για να οδηγήσουν όλη την στρατηγική ισότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια στρατηγική που πρέπει να συνδέεται με την κοινωνική ατζέντα, την νομοθεσία κατά των διακρίσεων και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο. Εμείς δεν θεωρούμε ότι μια στρατηγική θα πρέπει να δίνει μονάχα εντολές εκ των άνω προς τα κάτω, χωρίς να εφαρμόζεται σε εθνικό επίπεδο. Θα πρέπει να υπάρχει σαφή σύνδεση σε αυτά τα επίπεδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δει τρόπους να ξεπεράσει μια πατερναλιστική αντιμετώπιση στο να ενσωματωθεί η στρατηγική για τους Ρώμα σε όλες τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν πρέπει να ταινίζει τους Ρώμα ως παθητικούς αποδέκτες πολιτικής. Μέχρι τώρα είδαμε πολλά προβλήματα, προγράμματα στρατηγική σε εθνικό επίπεδο όπου οι πολιτικοί και οι κυβερνητικές αρχές δείχνουν καλή θέληση να κάνουν κάτι για τους Ρωμά, αλλά επειδή αλλά οι Ρωμά δεν έχουν εμπλακεί σχεδόν ποτέ στο σχεδιασμό και την εφαρμογή αυτών στρατηγικών, παραμένουν στη, στη θέση των παθητικών αποδεκτών, πολλές φορές ούτε καν αποδεκτών. και επιπλέον οι Ρωμά θα πρέπει να αναλάβουν και αυτοί οι ευθύνε και ένα ηγετικό ρόλο σε μια ευρύτερη στρατηγική ισότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα βοηθήσει όχι μόνο αυτού αλλά και όλη την ευρωπαϊκή κοινωνία. Η μειονεκτική θέση των Ρωμά στην Ευρώπη έχει και κοινωνικέ και πτυχέ και πτυχέ ταυτότητε. Δεν θα πρέπει οι στρατηγικέ να αντιμετωπίσουν την ε, κατάσταση των Ρώμα ούτε σε κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, ούτε σε εθνοτικό επίπεδο. Θα πρέπει να συνδεθούν οι δύο στόχοι της κοινωνικής ε, ενσωμάτωσης και του σεβασμού για την ταυτότητα των Ρωμά. Ε, σεβασμός των δικαιωμάτων τους είναι δυνατός μόνο αν καταλάβουμε ότι αυτά τα δύο στοιχεία είναι δύο, δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος. Για να έχουμε λοιπόν πλήρη και αποτελεσματική ισότητα για τους Ρώμα, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πλήρη προστασία των θεμελιωδών αστικών δικαιωμάτων των Ρωμά, μεταξύ των οποίων και μη διέκριση, ίση πρόσβαση, ίσες ευκαιρίες πρόσβαση σε εκπαίδευση ποιότητα. Γιατί όπως φάνηκε και από τι προτεραιο... τις προηγούμενες είπαν ορισμένοι ότι είναι σύμφωνα με το Σύνταγμα και τα έγγραφα ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλοι στο κράτο μα έχουν τα ίδια δικαιώματα. Μπορεί να έχουν τα ίδια δικαιώματα σε επιχάρτου, αλλά όπως λένε και οι αυτό μας ενδιαφέρει δεν είναι η τυπική ισότητα, αλλά η ουσιαστική ισότητα. Θέλουμε λοιπόν την, την ουσιαστική ισότητα στην πράξη. Έχουν πρόσβαση σε σχολεία οι Ρωμά, αλλά άμα αυτά τα σχολεία είναι χωριστά, αυτό δεν είναι θετικό. Βλέπετε ακριβώς πώς λειτουργούν τα χωριστά σχολεία όπου τα παιδιά 13-14 χρονών δεν έχουν ακόμα να μάθει να διαβάσουν και να γράφουν. Είναι απαραίτητο λοιπόν να υπογραμμίσουμε ότι δεν πρόκειται μονάχα για πρόσβαση στα σχολεία, αλλά πρόσβαση σε εκπαίδευση ποιότητος. Ίση πρόσβαση στην απασχόληση, ίσες ευκαιρίες να είναι αυτοαπασχολούμενοι, ίσες ευκαιρίες για στέγαση και υγειονομική περίθαλψη και πλήρη συμμετοχή με όλους τους άλλους στον οικονομικό και κοινωνικό στίβο. Επειδή έχει οριμάσει αρκετά το θέμα το Ρωμά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επειδή η εστίαση μόνο στα θέματα το Ρωμά μπορεί να έχουν αποτελέσματα μπούμεραγκ, η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να αποφύγει να διαχωρίσει πλήρως το θέμα το Ρωμά και να δημιουργήσει τελείως χωριστές δομές για τους Ρωμά. Αντίθετα, θα πρέπει να έχουμε μια δομή η οποία αν λειτουργήσει καλά μπορεί να είναι ένα υπόδειγμα για άλλες μειονεκτικές ομάδες και εθνοτικές ομάδες και μειονότητες όπου αυτό είναι απαραίτητο βέβαια γιατί υπάρχουν πολλά στοιχεία που δείχνουν ότι αν βασιστούμε μονάχα στις γενικές πρακτικές στον κύριο Κόρμο οι Ρωμά <clears throat> εξακολουθούν να είναι θύματα διάκρισης εξακολουθούν να είναι οι πιο μειονεκτικές κοινότητες στην κοινωνία στην οποία ζουν Πιστεύουμε λοιπόν ότι όταν και όπου αυτό είναι απαραίτητο θα πρέπει να υπάρξει μια πιο στοχευμένη προσέγγιση για αυτές τις πολιτικές. Να υπάρχουν πολιτικές ειδικά στοχευμένες στους Ρωμά, αλλά επί τη βάση των 10 βασικών αρχών που αναφέραμε προηγουμένως. Πιστεύουμε ότι αυτή η γενική πολιτική θα πρέπει να έχει μια ιδιαίτερη πτυχή για του Ρωμά. Προτεραιότητες στρατηγικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να εστιάσει σε μερικά κέρια θέματα τα οποία θα έχουν αποτέλεσμα βραχιών απόλαπλασιαστικό. Θεωρούμε ότι τα εξή σημεία μπορούν να είναι τέτοιε προτεραιότητε. Καταρχήν, αντιμετώπιση το, της νεαρής παιδικής ηλικία, όπως το αναφέραν και πολλοί άλλοι ομιλητέ, η μετάβαση από το σχολείο στην κερδοφόρα απασχόληση, αντιμετώπιση των ρατσιστικών στερεοτύπων και προκαταλήψεων. Πιστεύουμε ότι αυτές πρέπει να είναι οι τρεις διαστάσεις για τη μελλοντική μας στρατηγική για τους Ρωμά. Η καθεμία από αυτές τις προτεραιότητες θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με πλήρη τρόπο σε ό,τι αφορά την, ε, την παρουσία των εμπλεκομένων, των κύριων παικτών, των ε, αποδεκτών επίσης. Η πολιτική για την νεαρή ηλικία θα πρέπει να οδηγήσει σε μια συστημική αλλαγή η οποία θα επηρεάσει ένα αριθμό από αλληλένδετους τομείς για να εξασφαλίσει ότι υπάρχει ουσιαστική ισότητα των παιδιών των Ρωμά και των μη Ρωμά όταν μπαίνουν στο σχολείο. Αυτό σημαίνει υποστήριξη των οικογενειών, στέγαση και προσχολική εκπαίδευση. Υπάρχει ένα πολύ οξύ πρόβλημα της μη φίτησης των ε, παιδιών των Ρωμά στα σχολεία λόγω ένδυας. Αυτό πρέπει να είναι ένα κέριο θέμα, ένα κατεπήγον θέμα παρέμβασης. Εκεί πρέπει να εμπλακούν πολλαπλή φορείς και να αντιμετωπιστούν όλες οι πτυχές που έχουν να κάνουν με την κοινωνικοποίηση των παιδιών στη σχολική ηλικία. Και εφόσον μιλάμε για όλους αυτούς τους παράγοντες, θέλω να πω το εξή ότι μέχρι τώρα πάντα αντιμετωπίζουμε τους συνήθεις ύποπτους, δηλαδή τοπικές κυβερνήσεις, κεντρικές κυβερνήσεις και φορείς κοινωνία των πολιτών. Αλλά επειδή μιλάμε για δύο ε, διαστάσεις, για μη διάκριση και ε, κοινωνική συμπερίληψη, η Λίβια και η ομάδα της προτείνουν και μία ακόμα πτυχή, κοινωνικο-οικονομική αναβάθμιση της κοινότητας των Ρωμά. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μπουν και άλλοι παίκτες στο γήπεδο, όπως παραδείγματος χάρη οι επιχειρηματίες πρέπει και αυτοί να παίξουν κάποιο ρόλο στο, στην αναβάθμιση του κοινωνικονομικού επίπεδου των Ρωμά. Θα πρέπει να ξεπεράσουμε τα στερεότυπα και να αντιμετωπίσουμε τους Ρωμά ως ίσους και να αντιμετωπίσουμε τις προσεγγίσεις που είναι καθαρά φολκλωρικές. Να μπορούν λοιπόν να καταλάβουν και οι μη Ρώμα την κουλτούρα των Ρωμά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί πιστεύω ότι οι προκαταλήψεις βασίζονται στην έλλειψη πληροφόρησης. Η πληροφόρηση είναι η γνώση, είναι ένα από του καλύτερου τρόπου να αντιμετωπίσουμε τι προκαταλήψει. Αυτοί που είναι προκατελημένοι το κάνουν γιατί δεν ξέρουν πολλά πράγματα για του Ρωμά. Με τι πληροφορήσει, με την καλύτερη πληροφόρηση λοιπόν, νομίζω ότι όλα αυτά τα στοιχεία προκατάληψης μπορούν να εξαλειφθούν και έτσι <clears throat> να ξεπεραστούν και οι ρατσιστικές προσεγγίσεις. Όπω ελέγχεται επίση, η συμμετοχή των Ρωμά είναι σημαντική, θα πρέπει να είναι σαφώ καθορισμένη μέσα σε αυτή τη στρατηγική. Αυτή η στρατηγική θα πρέπει να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των Ρωμά σε όλα τα στάδια τη διαδικασία αυτή. Θα πρέπει να υπάρχουν σαφεί μηχανισμοί για ανταλλαγή απόψεων και διαβουλεύσει με του Ρωμά και οι στρατηγικέ αυτέ θα πρέπει να περιλάβουν στο δυνατόν περισσότερε απόψει. Η στρατηγική αυτή επίση θα πρέπει να ενθαρρύνει τα κάτι μέλη να αυξήσουν τη συμμετοχή των Ρωμά στη δημόσια ζωή, όχι απλώς κάθε τόσο καλούν σε μια ομάδα σκέψης και σε κάποιο συμβουλευτικό φορέα, αλλά να τους περιλαμβάνουν πλήρως και ενεργά στην δημόσια ζωή. Δεν είναι επαρκές να αντιμετωπίζουμε μονάχα το θέμα της απασχόλησης και της παιδείας, τα πολιτιστικά και κοινωνικά προβλήματα, χωρίς να εντοπίσουμε το πώς τέτοιες συνθήκες προκύπτουν από πολιτικές διακριτικού χαρακτήρα και πρακτικές διακριτικού χαρακτήρα. Και πάλι θέλω να υπογραμμίσω ότι και οι δύο προσεγγίσεις θα πρέπει να συνδυαστούν. Αν πάρουμε μονάχα την πτυχή της κοινωνικής συμπερίληψης και δεν έχουμε και την πτυχή της καταπολέμησης των διακρίσεων, ο κίνδυνος είναι ότι ίσως θα βελτιωθεί το επίπεδο το βιωτικό, αλλά θα είμαστε πάντα σε καταστάσεις ανθρώπων που δεν είναι φτωχοί πια, αλλά είναι απομονωμένοι και θύματα διακρίσεων, όπως αναφέρθηκε από προηγουμένους ομιλητές προηγουμένως. Αν όμως εστιάσουμε μόνο στην καταπολέμηση των διακρίσεων, <clears throat> θα έχουμε μια κοινότητα η οποία δεν αντιμετωπίζεται με διακριτικό τρόπο, αλλά θα ζει πάντα σε αποκλεισμό και σε ένδια. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι υπάρχουν υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτή τη στρατηγική για τις εθνικές, τοπικές και περιφερειακές αρχές. Κάθε αρχή θα πρέπει να υποχρεωθεί να πάρει με ενεργό τρόπο μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των Ρώμα και να υπάρχει επίσης και μία αξιολόγηση αντικτύπου για να εξασφαλίσουμε ώστε να αντιμετωπίσουν πλήρως τις υποχρεώσεις τους οι αρχές αυτές ε, τα θέματα αυτά και να υπάρχουν σαφείς οδηγίες και εντολές για να υπάρχει και αναθεώρηση και αξιολόγηση του ρόλου όλων των διοικητικών διατάξεων έναντι των Ρώμα. Οποιασδήποτε διατάξεις είναι διακριτικού χαρακτήρα θα πρέπει να τροποποιηθούν. Βέλτιστες πρακτικές δεν ξέρω αν έχουμε πολλές τέτοιες ευκαιρίες στην Ευρώπη, αλλά η Ιρλανδία και το Ενωμένο Βασίλειο ξεπερνούν και την θετική δράση. Πιστεύουμε ότι η θετική δράση είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να προωθήσουμε μια πραγματική ισότητα και να ξεπεραστεί η κατάσταση η μειονεκτική στην οποία βρίσκονται οι Ρωμά. Για τα θέματα ευθύνης. Όπως είπε ο Βαλέριο, η κυρία Ευθύνη θα πρέπει να είναι στους ώμους των κρατών μελών, γιατί εκεί λαμβάνουν χώρα όλα αυτά. Αλλά νομίζω ότι είναι μια διαμεμοιρασμένη ευθύνη, γιατί και οι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να συμμετάσχουν στην αντιμετώπιση όλων αυτών των προβλημάτων και στην ε, σχεδίαση και εφαρμογή της στρατηγικής. Αν το αφήσουμε μονάχα στα κράτη-μέλη, ο κίνδυνος είναι ότι οι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα έχουν καμία δυνατότητα ελέγχουν Ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν της αρέσει η έννοια του ελέγχου, αλλά όταν δίνουμε λεφτά πρέπει να ελέγχουμε πώς χρησιμοποιούνται αυτά τα χρήματα. Χρειάζεται λοιπόν μια καλύτερη σύνδεση με τις Εθνικές Αρχές και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός ο συντονισμός, για να το πω καλύτερα, πρέπει να υπάρχει και να είναι συνεχής. Και θέλω να κλείσω τώρα αν έχω ένα λεπτό ακόμα. Για την κρίση που αντιμετωπίζουμε. Εγώ ήμουν μέλος της ομάδος πρώτης γραμμής ούτως υπήν πριν από το 2000 που ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει σε νομοθεσία. Λέγανε πάντα τα ευρωπαϊκά όργανα ότι υπάρχει πάντα μια ατζέντα σε ό,τι αφορά την ισότητα και τα λοιπά και μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και στην περίπτωση των Ρωμά στο βαθμό που ενέπιπταν σε αυτή τη σφαίρα. Δεν ήθελε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει αυτή την ε, οδηγία κατά των διακρίσεων. Μετά από την κρίση που έλαβε χώρα στην Αυστρία το χειμώνα 1999-2000 και την άνοδο του εξτρεμιστικού δεξιού κόμματος στην εξουσία, είπε η Κομισιόν εντάξει θα καταθέσουμε μια οδηγία κατά των διακρίσεων, των ρατσιστικών διακρίσεων και ενεκρίθη. Σε επίπεδο στρατηγικής δεν υπήρξε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά οι τελευταίες κρίσεις, ιδίως στην Ιταλία και τη Γαλλία, έχουν παίξει ένα καταλητικό ρόλο για τις διαδικασίες αυτές και σήμερα πια μιλάμε για μια ευρωπαϊκή στρατηγική. Η ελπίδα μου είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα σκεφτούν συγκεκριμένα βήματα που πρέπει να αναλυθούν προς την κατεύθυνση αυτή, είτε θα είναι ένα πλαίσιο για τις εθνικές στρατηγικές ή μια ευρωπαϊκή ε, στρατηγική για τους Ρωμά, ρωμαϊκή στρατηγική, δεν έχει μεγάλη σημασία, αλλά όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν πριν έλθει και η επόμενη κρίση στο κεφάλι μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ιβανόφ. Σας ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας. Να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα τα θέματα που συζητήσαμε σήμερα. Φτάνουμε τώρα στο τελικό μέρος της απογευματινής μας συνεδρίασης, τη συζήτηση. Θα ήθελα να καλέσω όλους τους συμμετέχοντες να θέσουν τις ερωτήσεις τους και κατόπιν θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Γιαρούκα για να κλείσει την ακρόαση. Θα... Προς το παρόν η κυρία Λόχπιλάρ έχει ζητήσει το λόγο. Ρωτώ και άλλους εάν θέλουν να πάρουν το λόγο. Μετά από αυτό το τμήμα της συζήτησης. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είμαι μέλος της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, αλλά της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σήμερα το πρωί ζητήσαμε, τις, συζητήσαμε τις παραβιάσεις ε, των ανθρωπίνων ε, δικαιωμάτων στο Κωσυφοπαίδιο. Ε, επειδή όμως η Επιτροπή μας ε, δεν έχει όλες τις αρμοδιότητες. Ε, συζητάμε μόνο ε, το θέμα της παρεμβής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ που μου, δίνετε το, που μου δώσατε το δικαίωμα, να, που μου δώσατε τη δυνατότητα να, να ακούσω τη σημερινή παρουσίαση. Έχω μια ερώτηση προς τον κύριο Νι, ε, Νικολάη. Ε, είμαι από το Μόναχο. Θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ να έχω τα σχετικά έγγραφα, να ξέρω ποιος... Ε, ε ενέργησε και ποιος ε, αντέδρασε στην υπόθεση αυτή. Και έφτασα λίγο αργά, θα ήθελα όμως να αναφερθώ στην ορολογία. Θα ήθελα να συμφωνήσω με την Γερμανίδα συνάδελφο. Στο, στα πλαίσια της Γερμανίας η κοινότητα των Ρώμα επικρίνει όσους χρησιμοποιούν τον όρο ε, Μήπως τσιγκάνος, μήπως θα μπορούσε Προφανώς στις διάφορες χώρε λόγω τη διαφορετική ιστορία οι λέξεις χρησιμοποιούνται διαφορετικά. Θα πρέπει να σεβαστούμε αυτό που ζητάνε οι άνθρωποι αυτοί να αποκαλούνται στην κάθε χώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Περιμένω τον κατάλογο των ομιλητών που καταφτάνει. Υπάρχει άλλος που θέλει να πάρει το λόγο. Όχι. δύο άλλοι συμμετέχοντες, τον κύριο Μπάζ, παρακαλώ. Oui, je, ε, Θα ήθελα να παρέμβω ε, πάνω σε αυτό το θέμα για τους άτομα από το ξεφοπέδιο που έχουν απελαθεί ε, σήμερα. Είχαμε μια ανακοίνωση πάνω αυτό, αυτό το θέμα όχι μόνο πρέπει να μιλήσουμε για την κατάσταση των Ρώμα, καθώς και των ε, και αυτών των ανθρώπων που έχουν ε, ε, υπηκότητα σε, σε ευρωπαϊκό μέλος κράτος, αλλά και για τον τρίτον χρόνο τα άτομα. Υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν γεννηθεί στη Γερμανία, έχουν μεγαλώσει στη Γερμανία και σήμερα τι κάνουν, αντιμετωπίζουν την απειλή αυτή της απέλασης στο Κωσυβοπαίδιο. Ο Γκίντερ Γκράς, βραβείο Νομπέλ, πήρε θέση. Το διαδώσαμε αυτό, σε όλους τους, ε, κάναμε μια ανακοίνωση σε όλους τους Ευρωπαίους ε, Ευρωβουλευτές πάνω σε αυτό το θέμα, για να δείξουμε δηλαδή απλώς ότι το θέμα, θα επανέλθω από αυτό αύριο, ότι το θέμα ε, ενδιαφέρει πέρα από αυτά τα παράδειγματα που είχαμε πρόσφατο, αφορά πολλές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και όχι μόνο αυτές για τις οποίες σκέφτεται κανείς γενικά. I want to for, for, for the Θέλω να σας ευχαριστήσω για το, για το λόγο που μου δίνετε. Νομίζω τονίστηκε από πολλούς ότι όταν μιλάμε για στρατηγικές η ονομασία έχει σημασία. Από τη μία μεριά έχουμε μία έκκληση για, για, μια ευρωπαϊκή στρατηγική το Ρωμά και μια άλλη πρόταση από την Κομισιόν που έχει σαν τίτλο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο. Στο μέλλον, όταν καθοριστεί ακριβώς ο τίτλος, είναι απαραίτητο να εντοπίσουμε ακριβώς τι θέλει να επιτύχει αυτό το έγγραφο όταν λέω τι ακριβώς θέλει να επιτύχει, τι εκπροσωπεί, θα πρέπει και πάλι να ξεκαθαρίσουμε αν οι φορείς Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι κυβερνήσεις θέλουν να συμπεριλάβουν τους Ρώμα, αν θέλουν να τους εντάξουν ή αν θέλουν απλώς να βελτιώσουν την κατάσταση στο Ρώμα. Είναι δύο, τρία διαφορετικά πράγματα τα οποία πρέπει να κατανοήσουμε κάποια στιγμή. Γιατί το σχέδιο δράσης μιλάει για βελτίωση των συνδικών διαβίωσης στον Ρωμά. Λέει ακριβώς τι θέλει αυτό το σχέδιο. Ζητώ λοιπόν από τα μέλη του Κοινοβουλίου που είναι ακόμα παρόντα, στο μέλλον, στην έκθεσή σας, στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όταν ψηφίσετε, σας ζητώ να καθορίσετε τι ακριβώς θέλετε για να επανέλθω στο σχέδιο έκθεσης, στο σημείο υπαριθμών 2 θα προσκαλούσα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα τους πρότεινα ταπεινά, αντί να έχετε ένα μεγάλο κατάλογο ονίων στο κεφάλαιο 2, να έχετε υποκεφάλαια, υποεπικεφαλίδες να λέτε σε ποιες περιοχές θέλετε να δράσετε. Γιατί αυτός ο κατάλογος αν είναι τόσο μακροσκελής και εγώ ήμουν υπάλληλο τη Κομισιόν, δεν θα του έδινα σημασία. Είναι πάρα πολύ μακροσκελής αυτός ο κατάλογος, θα πρέπει τα πράγματα να τα οργανώσουμε σε μερικά μονάχα κεφάλαια. Τρίτο σημείο το οποίο θέλω να αναφέρω είναι το θέμα της συμπερίληψης των Ρώμα, το οποίο έχει αναφερθεί πολλές φορές στη συζήτηση που ξεκίνησε στις 3 η ώρα. Βλέπω σε αυτή την ίδια την αίθουσα να είναι ένα τεράστιο πρόβλημα στο κοινοβούλιο, στο πάνελ, στην ανάπτυξη στρατηγικής όπως είπε η Μιράντα. Ένα μεγάλο πρόβλημα, μια απουσία στα θεσμικά όργανα. Να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής μαζί σας, μέλη του κοινοβουλίου. Πέντε χρόνια δουλεύω, δούλεψα εδώ για ένα μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τότε ήμασταν μονάχα τρία άτομα που είχαν προέλευση Ρωμά. Τώρα υπάρχει μονάχα ένα άτομο και το θέμα είναι ακόμα πιο μεγάλο τώρα. Και το τελευταίο σημείο το οποίο θέλω να θίξω είναι περισσότερο ένα ερώτημα που θέλω να θέσω σε όλους. Πώς θα εξασφαλίσουμε ότι αυτή η στρατηγική θα εφαρμοστεί. Πώς εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει μια στεναρή πολιτική θέληση για την εφαρμογή αυτής της στρατηγικής. Είδαμε ότι Ακροδεξιοί πολιτικοί, η οποία είναι προφανώς εναντίον το Ρωμά. Και είναι πολλές φορές και αυτοί που παροτρύνουν να σκοτωθούν οι Ρωμά, να φωνευτούν οι Ρωμά, αυτοί βρίσκονται πολλές φορές μέσα σε κυβερνήσει. Νομίζετε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα υποστηρίξουν αύριο την υλοποίηση μιας στρατηγικής υπέρ των Ρώμα για τη βελτίωση της κατάστασή τους, για τη συμπερίληψή τους στην κοινωνία. Έχω πολλές αμφιβολίες. Γι' αυτό πιστεύω ότι στο μέλλον θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν έχουμε παραδείγματα αυτού του είδους και γι' αυτό θα πρέπει η Λίβια να εξασφαλιστεί ότι οι λέξεις τσιγκόινερ, ε, τσιγκάνι, τζίψις, όλα αυτά είναι ρατσιστικές ονομασίες και δεν μπορούν να περιλαμβάνονται εδώ. Ευχαριστώ. Ζητώ από όλου του ομιλητέ, αν θέλουν να αντιδράσουν, να πούνε κάτι. Κύριε Γκέντς, έχετε το λόγο. Νομίζω μπορούμε να συζητήσουμε τη συζήτηση αυτή για τα 15 λεπτά ακόμα. Θα ήθελα να σκεφτώ λιγάκι περισσότερο για αυτό που είπε ο κύριος Δεμιρόφσκι. Έχετε δίκιο ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε περί τίνος πρόκειται. όταν λέμε ότι δεχόμαστε την πρόταση της Κομισιόν για μια στρατηγική πλαισίου, εδώ το μήνυμα είναι ότι η πραγματική ένταξη και βελτίωση των συνθηκών ε, διαβίωσης των Ρωμά και αυτών που αγωνίζονται κατά των διακρίσεων θα πρέπει να συμβεί επιτοπίως στο τοπικό επίπεδο. Και από ό,τι ξέρω από τις προηγούμενες συζητήσεις έγινε σαφές ότι η Κομισιόν και γενικά οι φορεί της Ευρωπαϊκής Ένωση είχαν το φόβο ότι μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους Ρωμά θα έστελνε ένα μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα τα φροντίσει αυτά. Θα πάρει την ευθύνη απάνω της από τα κράτη-μέλη και τις τοπικές κοινότητες. Νομίζω ότι συμφωνούμε γενικά και θα ήθελα και τη δική σας άποψη ότι όπως προσπάθησα στη δική μου γνωμοδότηση, προσπάθησα να τονίσω και δεν ξέρω είδα τη γνωμοδότησή μου, να... Θα ήθελα να τονίσω ότι ο μόνος τρόπος να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα θα ήταν να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών επίπεδων. Όλα αυτά πρέπει να αντανακλώνται στο, στα εθνικά σχέδια ανάπτυξης, στη στρατηγική Ευρώπης 2020 κάτω από την επικεφαλίδα περιεκτική ανάπτυξη θα πρέπει να αντανακλώνται στα λειτουργικά προγράμματα, στα τοπικά σχέδια και στα πιο πολύπλοκα προγράμματα που έχουν να κάνουν με απασχόληση, με στέγαση κτλ. Αν δεν έχουμε τέτοιες εγκάρσιες μορφές συνεργασίας, δεν νομίζω ότι μπορεί να επιτεθεί τίποτα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε ότι μπορούμε να τα συζητάμε τα θέματα αυτά διαμακρών. Είχαμε πολύ ωραίες παρουσιάσεις και ομιλίες και συμφωνώ απόλυτα με αυτούς εξ ημών με ύψιλον ότι μιλήσαμε πολύ για τα θέματα αυτά, αλλά δεν είδαμε συγκεκριμένα εργαλεία για, για την υλοποίηση αυτών των στρατηγικών. Αυτό που προσπαθώ να κάνω στη γνωμοδότησή μου. Συζητούμε τώρα περισσότερο το πολιτικό στοιχείο και όχι το νομικό στοιχείο. Αυτό το οποίο προσπάθησα να κάνω είναι να καταλήξω σε συγκεκριμένες προτάσεις πώς να υπάρξουν εξαρτήσεις και προϋποθέσεις για τη χρήση των ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς να υπάρξει μια εγκάρσια προσέγγιση, ώστε παντού να υπάρχουν οι ίδιοι στόχοι, να υπάρχουν στοιχεία για βαθμονόμηση. των να υπάρχουν έρευνε που μα λένε τι γίνεται, ποιο επηρεάζεται, ποιο δεν επηρεάζεται από όλα αυτά τα προγράμματα. Να μπορέσει όλο ο μηχανισμό λήψη απόφαση να είναι κοντύτερα στα μέλη των κοινοτήτων αυτών και στα κράτη-μέλη. Αν οι αποφάσει λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κανεί δεν θα μπορέσει να υποστηρίξει τι σημαντικέ μικρέ τοπικέ ε, πρωτοβουλίε αρκετά ώστε να μπορέσουν να αναπτυχθούν και να δώσουν αποτελέσματα. Και αν δεν έχουμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, και αυτό που άκουσα από τις παρουσιάσεις σας, από το Φορέα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων κτλ. Νομίζω ότι ήταν τέτοιου είδους συγκεκριμένες προτάσεις. Ξέρουμε τι θα θέλαμε να έχουμε σαν αποτέλεσμα στο τέλος, αλλά δεν ξέρουμε πώς να το επιτύχουμε και νομίζω ότι πρέπει να επεξεργαστούμε όλα αυτά τα θέματα στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Υπάρχει άλλος που θέλει να πάρει το λόγο. Εάν όχι, να δώσω το λόγο στην κυρία Γιάρουκα για να κλείσει τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ όλους για τη συνεισφορά σας. Ίσως οι τελευταίες ερωτήσεις να ήταν οι πιο αποκαλυπτικές διότι η ακρόαση αυτή στόχο είχε να συζητήσουμε τι είδους ε, στρατηγική, ευρωπαϊκή στρατηγική θέλουμε για τους Ρώμα και πώς ε, η Κομισιόν μπορεί να προετοιμαστεί ε, για την εκπόνηση του νέου εγγράφου τη και πώς μπορούμε να φροντίσουμε τότε να καταλήξουμε σε ένα σχέδιο δράση. και να ε, είμαστε βέβαιοι ότι στις 26 Ιουνίου όλα τα κράτη-μέλη θα υπογράψουν την ε, κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική. Βλέπουμε όμως τη συζήτηση στην οποία συνέβαλαν ε, και οι μη κυβερνητικέ οργανώσει και όλοι οι φορεί Όλα αυτά είχαν να κάνουν με το μικρό, το στενό μονοπάτι ε, που θα μας οδηγήσει στην επιτυχία. Κάποιες χώρες δεν είναι έτοιμες να υπογράψουν. Έχουμε κοιτάξει όλες ε, τις ευρωπαϊκές ε, συνθήκες. Έχουμε 62 εκτιμώντας στο έγγραφο αυτό που να έχουν να κάνουν με τις προϋποθέσεις για να ε, πραγματοποιηθεί μια στρατηγική. Τώρα λοιπόν για πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή πολιτική ε, βρισκόμαστε σε θέση όπου ε, να μπορεί να εγκριθεί μια τέτοια στρατηγική. Η έκθεση αυτή έχει υποβληθεί στην Επιτροπή μας πριν κάποιες μέρες. Ακούσαμε πολύ καλές γνωμοδοτήσεις από τέσσερα κράτη-μέλη. Όλα αυτά δείχνουν το πώς Μπορεί να έχουμε, μπορούμε να έχουμε ευρωπαϊκή στρατηγική για τους Ρώμα που να δεσμεύει όλα τα κράτη-μέλη διότι υπάρχει ήδη η νομική βάση, έτσι δεν είναι. Δεν χρειαζόμαστε πολλά λοιπόν. Πρέπει τα κράτη-μέλη να συμμορφωθούν με ε, τις υποσχέσεις τους και με τα καθήκοντα, ε, τις αρμοδιότητες που τους δίδονται μέσω των ε, όλων των συνθήκων με τις ευρωπαϊκές στρατηγικές που ήδη έχουν εγκριθεί. Τώρα πια λοιπόν πρέπει να φροντίσουμε από την ε, βάση, από τους ε, δημάρχους μέχρι το ευρωπαϊκό επίπεδο ε, να μπορεί να εφαρμοστεί η στρατηγική. Μιλάμε για μη διάκριση, μιλάμε για ίσες ευκαιρίες όσον αφορά την απασχόληση και την εκπαίδευση. Και όλοι γνωρίζουμε ότι με το καλό αυτό σύστημα παρακολούθησης ε, κανένα κράτος μέλος δεν θα παραβιάσει τη στρατηγική αυτή, διότι χάνουν ψήφους. Μάλλον τα τελευταία 20 χρόνια δεν, δεν κάναν τίποτα τα κράτη-μέλη για να μην χάσουν ψήφους. Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή στρατηγική για τους Ρώμα, νομικά δεσμευτική, Βλέπω ότι υπάρχουν οι απαραίτητε δομέ. βλέπω ότι υπάρχουν ε, τα απαραίτητα χρήματα, το λέω αυτό και στην έκθεσή μου. Νομίζω ότι γίνεται διαβούλευση εδώ και πολλά χρόνια ε, με τόσους διαφορετικούς ανθρώπους, με τόσες ε, κυβερνήσεις. Πιστεύω λοιπόν ότι όλα αυτά είναι δυνατά. Μόνο και μόνο για το λόγο ότι οι Ούγγροι είναι διατεθειμένοι να πολεμήσουν, να αγωνιστούν για το θέμα αυτό. Κανένα άλλο κράτο μέλο δεν είπε ότι διαθέτει για μια στρατηγική για τους Ρώμα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν μια έκθεση πρωτοβουλίας μπορεί να αποτελέσει ε, την βάση για ένα κοινοτικό σχέδιο δράσης και πιστεύω ότι ο ρόλος του Κοινοβουλίου ε, είναι να σπρώξουμε την ε, Επιτροπή προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα πρέπει να βεβαιωθούμε Ε, ότι όλα τα κράτη-μέλη που ε, εκπροσωπούνται εδώ πέρα και που πριν πέντε χρόνια ε, τόσο ευχαρίστως υπέγραψαν την άχρηστη, το, το άχρηστο ψήφισμα για τους Ρώμα, όλοι αυτοί λοιπόν τώρα να συμμετάσχουν, να συμμορφωθούν όλα τα κράτη-μέλη που ε, ε, ε, υποβάλλουν λίγο ύποπτα δεδομένα προς την Επιτροπή, όλοι αυτοί θα πρέπει να, να συμμορφωθούν, θα πρέπει να φροντίσουμε τα χρήματα να φτάνουν όχι μόνο στους Ρώμα, σε όλους στην Ευρώπη που ζουν σαν τους Ρώμα, των οποίων το πρόσωπο σήμερα στην Ευρώπη είναι η Ρώμα. Αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι μιλάμε για έναν χάρτη κρίση για, τους, για όλους τους φτωχούς που ζουν σαν τους Ρώμα, διότι πιστεύω ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος να λύσουμε το πρόβλημα και να ξεπεράσουμε τα τελευταία 20 χρόνια αποτυχιών, όπου δεν υπήρχε καμία βούληση από πλευρά των πολιτικών. Ε, η Ευρώπη και η Κομισιόν κλείνανε ε, τα μάτια και το Συμβούλιο χαμογελούσε ευχάριστα που δεν χρειαζόταν να κάνει τίποτα. Και δεν, ε, σας τα ανέφερα όλα αυτά, δεν σας έχω καν αναφέρει το τι νιώθουν οι Ρώμα για όλα αυτά. Πιστεύω λοιπόν ότι η σημερινή μέρα είναι πολύ καλή ευκαιρία και θα ήθελα πολύ να είχα ακούσει πολύ περισσότερα σχετικά με το περιεχόμενο του εγγράφου αυτού που είναι γεμάτο από προτάσεις. Η Κομισιόν πολύ ευχαρίστω θα παραβλέψει τις προτάσεις αυτές εφόσον δεν ακούγονται αρκετά δυνατά. Ε, Στόχο μας είναι λοιπόν να υψώσουμε τη φωνή μας ώστε να φροντίσουμε να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία αυτή στο επακρόν. Ή τώρα ή ποτέ. Και με αυτό το πνεύμα ετοίμασα το συγκεκριμένο έγγραφο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Ολιβία. Σε υποστηρίζουμε σε αυτόν τον αγώνα. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές του απογεύματος όλες τις ε, ιδέες που μας ε, δώσατε. Θα συνεχίσουμε την ακρόαση αύριο το πρωί. Ξεκινούμε στις 9. Και νομίζω ότι θα έχει τόσο ενδιαφέρον όσο και στο πρώτο μισό του απογεύματος με τη συμμετοχή πολλών μελών και πολλών ομιλητών. Καλό βράδυ λοιπόν, καλή ξεκούραση και θα συνεχίσουμε αύριο σε 9 η ώρα αν θέλει ο Θεός στην ίδια του. Και ευχαριστούμε τα κορίτσια που μεταφράζουν.